gentlemen, Υπάρχουν άδεια καθίσματα ακόμα στην αίθουσα. Δεν έχουμε πάρα πολλούς ε, παρόντες μέσα στην αίθουσα, είναι αλήθεια. αλλά ακόμα και αν κάποιοι συνάδελφοι δεν είναι παρόντες, νομίζω ότι εμείς, ε, ε, εφόσον μάλιστα εργαζόμαστε σε web streaming, οφείλουμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο σημείο στην ημερησία διάταξη είναι η έγκρισή της. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για την ημερήσια διάταξη. ή Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Συνεπώς θα ήθελα να σας ζητήσω να εγκρίνετε τα πρακτικά πλέον των συνεδριάσεων της 18ης Δεκεμβρίου, 22ης Ιανουαρίου, 11ης Φεβρουαρίου και 24ης Φεβρουαρίου. αν δεν έχετε παρατηρήσεις ε, για τα πρακτικά. Υποθέτω ότι θεωρούνται δεκτά. Τώρα, ανακοινώσει της Προέδρου, της κυρίας Χιούμπνερ, της πραγματικής Προέδρου, θα έρθει αργότερα. Εγώ δεν έχω κάτι να πω εδώ. Και έτσι πηγαίνουμε απευθείας στο βασικό θέμα την εξωτερική μελέτη την οποία ζητήσαμε εμείς για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μία μελέτη η οποία δεν έχει φτάσει στην τελική της φάση ακόμα, αλλά θα θέλαμε, έστω και στην παρούσα φάση, να δούμε πού βρίσκεται η συζήτηση. Και θα ήθελα να ζητήσω από την παρουσιάστρια της ομιλίας να πάρει το λόγο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και μια ανταλλαγή απόψεων. Έχει το λόγο λοιπόν η κυρία Σιμώνα Μίλιο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας εδώ σήμερα για να παρουσιάσουμε την πρόοδο της εργασίας μας, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Καταρχάς θα παρουσιάσω το πλαίσιο στο οποίο έγινε η μελέτη, το πώς βλέπουμε εμείς την κρίση, τα βασικά ευρήματα τα οποία τα έχουμε διαιρέσει σε ποσοτικά ευρήματα και κατά περίπτωση μελέτες και κάποιες ε, ε, παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική συνοχή ανταποκρίθηκε. Το πλαίσιο της μελέτης τώρα. Το πλαίσιο της μελέτης λοιπόν εξελίσσεται, αναπτύσσεται είναι μια κρίση η οποία εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. <clears throat> Έχει χτυπήσει, αν θέλετε, την Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά σκληρά. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4% και η βιομηχανική παραγωγή κατά 20% από το 2009. Το 2008 ξεκίνησε το πρόγραμμα ανάκαμψης για συντονισμό της δράσης μείωσε τις επιπτώσεις στο πρόγραμμα αυτό τις συνέπειες της κρίσης αλλά ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί ότι πράγματι ε, μπόρεσαν οι περιφέρειες να προσαρμοστούν. Στόχος της μελέτης καταρχάς ήταν να αξιολογήσουμε σε ποσοπτικό επίπεδο και αναλυτικό επίπεδο τις επιπτώσεις σε οικονομικό, κοινωνικό και εδαφικό επίπεδο και δεύτερον να δούμε τις απαντήσεις της πολιτικής συνοχής. Ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε εμείς είναι ότι η κρίση εξελίσθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη ξεκίνησε το 2008, είναι η λεγόμενη κρίση του ιδιωτικού χρέους και μετά μετετράπη σε δημόσιο χρέος. Η κρίση του ιδιωτικού ε, χρέους αφορά τρεις τομείς, την παραγωγή, τις κατασκευές και τα χρηματοπιστωτικά. Ε, φυσικά κάθε μία από αυτές τις κρίσεις χτύπησε διαφορετικές περιπτώσεις. Αν δούμε την πρώτη φάση του ιδιωτικού χρέους, της κρίσης του ιδιωτικού χρέους, βλέπουμε ότι χτυπήθηκαν καταρχάς ε, μέσω της μείωσης της βιονικής παραγωγής οι βιομηχανικές περιοχές χώρες του Βορρά, Ηνωμένο Βασίλειο, κάποιες περιοχές των ανατολικών χωρών, ο βορράς της Ιταλίας, η κεντρική Αυστρία και ο νότος της Γερμανίας. Ταυτόχρονα ο τομέας των κατασκευών της οικοδομής ε, λειτουργήσε διαφορετικά, είναι πιο ελαστικός στην σφαιρική ζήτηση και συνδέεται περισσότερο με τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Ο τομέας των κατασκευών λοιπόν που επηρέασε ε, κάποιες χώρες πιο σημαντικά από άλλες, ε, τη Βαλτική, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και τη Μεσόγειο γενικότερα. Και τέλος ο χρηματοπιστωτικός τομέας <coughs> χτύπησε κυρίως τις πρωτεύουσες όπου υπάρχουν ε, μεγάλες παρουσίες πιστοτικών ιδρυμάτων, χρηματιστηρίων κτλ και μετετράπη σε φράση δημοσίου χρέους. Ε, η κρίση αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από διάφορους παράδοντες όπως η μείωση των φορολογικών εσόδων, μείωση κοινωνικών επενδύσεων, έλλειψη πιστώσεων, υψηλό κόστος δανεισμού και αυτό χειροτέρευσε και με την εισαγωγή μέτρων λιτότητας. Έτσι βλέπουμε το πώς παρουσιάζεται η κρίση λοιπόν. Τώρα προσπαθούμε να δούμε ε, τα κανάλια μεταφοράς, τους διάβλους μεταφοράς της κρίσης, πώς ε, πέρασε στο εθνικό επίπεδο η κρίση και από το εθνικό στο διεθνές. Καταρχάς, διαθεσιμότητα πιστοτική, επιτόκια, εμπόριο και ε, ζήτηση εσωτερική και τοπική. Αυτή τη στιγμή εντοπίσαμε τους κανόνες αυτούς, προσπαθούσαμε να δούμε πώς αυτό το εθνικό επίπεδο ανταποκρίθηκε στα προβλήματα που έθεσε η κρίση και αυτό ονομάζουμε εμείς περιφερειακά συστήματα αντοχής. Ε, ανάλογα με τις περιφέρειες προσπάθησαν να αντέξουν τις επιθέσεις λόγω της κρίσης. Τρεις διαστάσεις εδώ. Καταρχάς, εξειδίκευση περιφερειακή, ανθρώπινη πόρη και ε, καινοτομία. Περνώντας τώρα στην ποσοτική ανάλυση και στην ανάλυση των μεμονωμένων περιπτώσεων. Καταρχάς προσπαθήσαμε να δούμε αν συνδέονται οι παράγοντες ε, της ε, μετάδοσης της κρίσης με τους παράγοντες αντοχής απέναντι στην κρίση. Η ανάλυση των επιμέρους περιπτώσεων είναι μια ε, ποσοτική ανάλυση μέσω, ε, η οποία έγινε μέσω συνεντεύξεων. Λοιπόν, η ποσοτική ανάλυση βρίσκει τρία βασικά θέματα. Πρώτον, αυτό που ονομάζουμε North-South Metaphors, δηλαδή Δύο ε, βασικά χαρακτηριστικά εδώ έχουμε ε, επίσης και το σύνδεσμο ανάμεσα στις οικονομικές συνθήκες προκρίσεως και τις επιπτώσεις της ύφεσης. Αυτές ε, οι metaphors, λέει ο Μιλήτρια, δεν μπορούν να δείξουν ποιο είναι το περιεχόμενο ακριβώς της κρίσης. Ο υπηρετικός τομέας επηρεάστηκε πολύ λιγότερο από τις περιφερικές χώρες στο εξωτερικό του κοινοτικού κύκλου δηλαδή. Οι χώρες που ε, φύγησαν λιγότερο είναι η Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία, ενώ περιφερικές ζώνες χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, τμήματα της Ελλάδας, Ελλάδα, Κύπρος, Λιθουανία, Λετωνία και Εσθονία. Καταρχάς υπάρχουν δύο αντιτιθέμενες εδώ αντιφατικές τάσεις. Βλέπουμε ότι ε, γενικά σε κάποιες χώρες υπάρχει ισχυρή απάντηση αλλά αντοχή. Γενικά το πρόβλημα παραμένει. και θα πρέπει να δούμε και το σύνδεσμο ανάμεσα στις οικονομικές συνθήκες ε, προκρίσεως και τις επιπτώσεις της ε, ύφεσης. Οκτώ παραμέτρους επιλέξαμε εμπειρικά. Τέσσερις για οικονομικά επίπεδα, δύο παραμέτρους για θέματα κοινωνικά και δύο παραμέτρους για ε, θέματα εδαφικής και περιφερειακής συνοχής στον τομέα των υποδομών κυρίως. Εξετάσαμε τις παραμέτρους αυτές ε, σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από την κρίση και μετά την κρίση και είδαμε ότι κάποιοι από αυτούς συνδέονται πράγματα με τις επιπτώσεις άμεσα της κρίσης. Σχετικά με τους παράγοντες αντοχής, αν θέλετε, ανθεκτικότητας. Εμείς εξετάσαμε τους ανθρώπινους πόρους, είδαμε ότι οι, ο, ανθρώπινοι πόροι και η καινοτομία δεν συνδέονται άμεσα με τις οικονομικές επιδόσεις κάθε περιοχής. Και αυτό γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι κάποιες επιπτώσεις βραχυπρόθεσμες ενώ συνδέεται ε, το φαινόμενο αυτό με την μακροπρόθεσμη περισσότερο οικονομική ανάπτυξη. Σχετικά με το δεύτερο τμήμα της μελέτης αυτής, τις περιπτωσιακές έρευνες, επιλέξαμε τέσσερις χώρες, Πολωνία, Βουλγαρία, Ιταλία και Γερμανία ακριβώς λόγω του διαφορετικού επίπεδου με το οποίο εφήγησαν. Σε αυτές τις χώρες επιλέξαμε δύο περιοχές, δύο περιοχές σύγκληση στην Πολωνία, δύο περιοχές στην Ιταλία όπως η Καμπανία, δύο περιοχές σύγκληση στη Γερμανία και δύο ε, περιφέρειες στη Βουλγαρία η βορειοανατολική και η νοτιοδυτική. Αυτό μας επέτρεψε να συλλέξουμε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούσαμε για τις περιφερειακές διακυμάνσεις. Τα βασικά ευρήματα αυτών των επιμέρους αναλύσεων που έγιναν με, ε, όχι μόνο με δεδομένα, με συλλογή δεδομένων αλλά και με ε, συνεντεύξεις είναι ότι η Ιταλία μας δείχνει πώς γίνονται τα πράγματα Πώς δηλαδή η κρίση του ιδιωτικού χρέους έγινε κρίση δημοσίου χρέους. Αυτό στην αρχή δημιούργησε προβλήματα ανισότητας, οι βόρειες περιοχές στην αρχή εφήγησαν περισσότερο από τις νόητιες, αλλά τελικά είναι οι περιοχές αυτές οι οποίες ανέκτησαν θα έλεγα τη δύναμή τους ταχύτερα από ό,τι στο νότο. Στην Γερμανία, εκεί ε, υπήρξε η εμπειρία της κρίσης από τις αρχές του 2009, υπήρξε μια ισχυρή ανάκαμψη λόγω του εμπορίου με τις μη κοινοτικέ αγορές. Η ανάκαμψη αυτή ε, επιταχύνθηκε επίσης και από την καινοτομία και τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού πάνω από τον κοινοτικό ε, μέσο όρο για την Πολωνία. Εδώ έχουμε μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με πιο αναπτυγμένες οικονομίες. Βλέπουμε ότι τα πιστοτικά ιδρύματα δεν υπέφεραν ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της, αγοράς, της κατάπτωσης της αγοράς ομολόγων στη ΣΥΠΑ. Η πολωνική οικονομία εξαρτάται λιγότερο από τις εξαγωγές, εποφελήθηκε από την απομείωση του πολωνικού σλότη, και αντίθετα με άλλες και κυβερνήσεις η πολωνική κυβέρνηση μείωσε τους φόρους για να αυξήσει την εσωτερική κατανάλωση. Όλα αυτά στήριξαν λοιπόν την Πολωνία. Και η τελευταία χώρα την οποία μελετήσαμε ήταν η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία είναι ένα παράδειγμα το οποίο έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με την λεγόμενη περιφερειακή η εδαφική διάσταση αν θέλετε. Είδαμε επίσης και τα μεθοριακά προγράμματα, τα διαμεθοριακά προγράμματα για να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο περιφερειακής συνοχής. Η βουλγαρική οικονομία διασυνδέεται στένα με τους εμπορικούς εταίρους και έτσι η Βουλγαρία ε, ε, έζωσε την κρίση και σε εσωτερικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εμπορικών συναλλαγών με τις γειτονικές χώρες. Η μεταφορά της κρίσης λοιπόν στην Βουλγαρία ανταποκρίνεται στην πορεία την οποία είδαμε στην αρχή. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην Βουλγαρία βέβαια εξακολουθεί να έχει κάποια θέματα. <clears throat> Τώρα τι απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε η κρίση οδήγησε σε δύο βασικές επιπτώσεις σε σχέση με την πολιτική συνοχής. Καταρχάς αλλαγή της εφαρμογής των πολιτικών μας, εφαρμόστηκαν οι αλλαγές έτσι ώστε να βελτιωθούν η απορροφητικότητα και οι τοπικές δυνατότητες. Έπρεπε να διατηρήσουμε επίσης και ένα ικανό επίπεδο επένδυσης αυτό φαίνεται από την ανάλυση την οποία κάναμε και από τις συνεντεύξεις τις οποίες κάναμε στις διάφορες χώρες μέλη. Όλοι συμφώνησαν λέγοντας ότι η πολιτική συνοχή είναι ε, θεμελιώδης για να διατηρηθούν τα επίπεδα επενδύσεων, ιδιαίτερα στις χώρες όπου οι δαπάνες αυτές ήταν υψηλές, οι ανάγκες ήταν υψηλές. Ταυτόχρονα προσπαθήσαν να αποφύγουν μια κλιμάκωση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, ιδιαίτερα στις περιοχές σύγκλησης όπως η Ιταλία, δύο Ιταλικές περιοχές, δύο Πολωνικές περιοχές. Έγιναν αλλαγές με δύο τρόπους βασικά, έτσι ώστε να προσαρμοστεί η αρχική στρατηγική στις νέες αλλαγές και στα νέα σενάρια. Πρώτον, υπήρξε μια μεταφορά θα έλεγα από τις μακροπρόθεσμες προοπτικές που είχαν τεθεί στην αρχή και αυτό είναι λογικό γιατί η πολιτική συνοχή ανταποκρίνεται και συγκεντρώνεται στις άμεσες ανάγκες. Δεν έχει νόημα βέβαια από την άλλη να στηρίζουμε τις άμεσες ανάγκες και να αποτυγχάνουμε στις μαθοπρόθεσμες προοπτικές ιδιαίτερα στον τομέα των δημοσίων δαπανών. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ε, η περιφερειακή πολιτική δεν λειτουργήσε σαν ένας επιπλέον πόρος αλλά στην ουσία αντικατέστησε από όλες τέντες πόρους. Υπήρξε καθυστέρηση λοιπόν και στην ανταπόκριση στην κρίση, υπήρξε απλούστευση γενικά ε, και της εφαρμογή των μέτρων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης, ιδιαίτερα μέσω του θέματος της συγχρηματοδότησης. Βέβαια αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Βασική στρατηγική ήταν να απλοποιηθεί ε, η διαδικασία συγχρηματοδότησης για να μην χειροτερεύσει η κατάσταση για τις επιχειρήσεις και τις τοπικές αρχές. Υπήρξαν επίσης και κοινέ απαντήσεις στον τομέα της πολιτικής συνοχής στις περιοχές συνοχής σύγκλησης. Μάλλον είδαμε ότι υπήρξαν περιφέρειες οι οποίες προσπάθησαν να αυξήσουν με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο την απορροφητικότητά τους. Ταυτόχρονα σε άλλες περιοχές άλλαξε η στρατηγική τους σε επίπεδο διαχείρισης, όχι όμως σε επίπεδο στόχων. Έτσι οι περιφέρειες οι οποίες είναι σε επίπεδο σύγκλησης χρησιμοποιούν την πολιτική συνοχής για να αντιμετωπίσουν τα θέματα τα αναπτυξιακά με μια στρατηγική η οποία δεν έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Η πολιτική συνοχής λοιπόν φαίνεται ότι δεν έχει ανταποκριθεί πλήρως γιατί στον τομέα της ανταγωνιστικότητας οι πολιτικές συνοχής ασχολήθηκαν με επιμέρους, με μικρά προβλήματα και όχι με μακροπρόθεσμα συνολικότερα θέματα. Και βλέπουμε στην γερμανική περίπτωση <clears throat> όπου έχουμε τις τοπικές, τα τοπικά χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας τα οποία επιτρέπουν τη μετρίαση των συνεπειών της κρίσης. Είδαμε επίσης στην περίπτωση της Βουλγαρίας και τα διαμαθοριακά θέματα. Καταρχάς βλέπουμε ότι σε επίπεδο διαμεθοριακών προγραμμάτων έχουμε χαμηλότερους πόρους λόγω μικρότερων ποσών που περνούν από τα διαφθορτικά ταμεία. Δεύτερον έχουμε ένα συγκεντρωτικό σύστημα το οποίο δεν επιτρέπει σε εύκαμπτη ανταπόκριση στις ανάγκες και τρίτον τα προγράμματα αυτά προσπαθούν να βελτιώσουν τις σχέσεις ανάμεσα στους τοπικούς πληθυσμούς, ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και θα πρέπει να εξεταστούν και σε σχέση με την επιτυχία τους σε αυτό το επίπεδο. Συμπερασματικά αυτό το οποίο φαίνεται εδώ και αυτό φαίνεται και από την ποσοτική ανάλυση είναι ότι στο μέλλον τα προγράμματα συνοχής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες εντατικότητας που διαφοροποιούνται γεωγραφικά και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όλες οι περιφέρειες με τον ίδιο τρόπο. Δεύτερον, είναι σαφές ότι οι περιφέρειες αντιμετώπισαν με διαφορετικό τρόπο την κρίση. Αυτό το οποίο έχει σημασία και είναι μια επιπλέον παρατήρηση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευέλικτη αντιμετώπιση, είναι όμως απαραίτητο να υπάρχει μια έννοια υπολόγου αν θέλετε, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα η δυνατότητα ελέγχου σωστού. Κάποια άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι οι διαφορές και η ισορροπία ανάλογα σε αυτό που ονομάζουμε soft outcome και hard outcome. Δηλαδή το soft outcome αφορά τα θέματα της απασχόλησης, τα ποσοστά απασχόλησης, τα θέματα της εμπιστοσύνης, τα οποία δεν εξετάσαμε σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Ενώ τα hard outcomes είναι δεδομένα αριθμητικά τα οποία αφορούν αυτούς οι οποίοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας μέσω της παρέμβασης των διαφορετικών ταμείων. Το τρίτο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η πολιτική σύνοχης προσπάθησε να ανταποκριθεί στην κρίση, υπήρξε μια ευθυγράμμιση ανάμεσα στα τρία βασικά ταμεία, τα περιφερειακά ταμεία, το κοινωνικό ταμείο και το ταμείο συνοχής. Υπήρξε ένα σωστό συντονισμός ανάμεσα στα τρία αυτά ταμεία και αν δούμε από τη μία την ε, ευθυγράμμιση των διαρθρωτικών ταμείων από τη μία και των υπολείπων από την άλλη θα δούμε ότι υπήρξε παράλληλη προσπάθεια. Ε, Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Είναι μία μελέτη αυτή η οποία παρουσιάζεται στο ενδιάμεσο διάστημα διότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα τώρα στα μέλη να σχολιάσω, να παρατηρήσω. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία στην ανάλυση σας. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Ωραία, εντάξει. Το πρώτο στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι ότι αναφέρεστε στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό ε, Πρόγραμμα Ανάκαμψης οικονομικής ανάκαμψης και δεν αναφέρεται καθόλου τα αποτελέσματα, το αποτέλεσμα εγώ πιστεύω ότι αυτά τα οποία αναφέρεται στην πολιτική συνοχή είναι λάθος, διότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 6 ε, εκατομμυρίων ευρώ προήλθε από το απόθεμα ε, του Ταμείου συνοχή 6 ε, δισεκατομμύρια ευρώ και δαπανήθηκε όχι για πολιτικέ συνοχή, αλλά δαπανήθηκαν αυτά τα 5,6 δισεκατομμύρια σε προγράμματα τεχνολογίας, σε προγράμματα πληροφορικής και το 2014 ζητήσαμε πολλές φορές από την Κομισιόν να μας εξηγήσει πώς αυτό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης έχει υλοποιηθεί, διότι έχει τελειώσει, ολοκληρώθηκε τις 31 Δεκάτου του 2013, δεν υπάρχει ούτε συν ένα ούτε συν δύο. Και θέλαμε να ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις, τι υλοποιήθηκε από το πρόγραμμα αυτό. Εσείς βασίσατε την ανάλυση σας στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, του υπάρχοντος, διότι αυτά τα οποία αναφέρεται είναι εντελώς εσφαλμένα. Δεν έχει τίποτα να κάνει με την πολιτική συνοχή. Απλώς χρησιμοποιήθηκαν τα αποθέματα από το Ταμείο Συνοχής και διοχετεύτηκαν σε τρεις ε, χρηματοδοτικές ε, πτυχές. Επίσης, με εντυπωσιάζει, εκπλήσωμε ιδιαίτερα που δεν έχετε προσέξει και αναφέρει διόλου τις διαφορετικές ε, προσεγγίσεις των κρατών μελών και αντιμετωπίσεις των κρατών μελών όσον αφορά την, την προσθετικότητα. Όπως ξέρετε η προσθετικότητα είναι υποχρέωση των κρατών μελών και ε, δημόσια, δημόσια συγχρηματοδότηση ε, πρέπει να συνάδει και να συντρέχει με την ευρωπαϊκή ε, συγχρηματοδότηση. Οι χώρες έχουν λοιπόν στην προσθετικότητα αντιδράσει πολύ διαφορετικά. Η Πολωνία την αύξησε 56%. Ε, η Ιταλία και η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ελλάδα την μείωσαν περίπου 22-23% ε, και αυτό δείχνει ότι πέραν της συγχρηματοδότησης οι χώρες αντιμετώπισαν τελείως διαφορετικά την προσθετικότητα, δηλαδή τις δημόσιες επενδύσεις. Αυτό είναι ένα σοβαρό στοιχείο και λείπει από την ανάλυση που κάνατε. Και τέλος, δεν καταλαβαίνω διόλου τη φιλοσοφία των ε, συμπερασμάτων σας. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο περισσότερο τι σημαίνει το soft outcome έναντι του hard outcome. Δεν καταλαβαίνω διόλου τι λέει αυτό. Ίσως άλλοι συνάδελφοι το κατανοούν, αλλά αυτό έχει γραφεί με τέτοια φιλοσοφική διάθεση που δεν καταλαβαίνω το βαθύτερο νόημα. Δηλαδή, αν μπορείτε πιο απλά να με εξηγήσετε τι σημαίνουν αυτοί οι δύο όροι, soft και hard outcome, διότι είναι μια σοβαρή μελέτη αυτή, μην γελιόμαστε. Ο πρόεδρος. Ε, ε, ε, ευχαριστώ, λέει ο κύριος Νίλσον. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, προέρχομαι από τη Σουηδία όπως ξέρετε και κατανοώ ότι υπάρχουν περιφέρειες στην Σουηδία που δεν μπορούν να συγκριθούν με περιφέρειες της Γερμανίας σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης. Και ε, πιστεύω ότι είναι καλό να υπάρχει μια τέτοια μελέτη στα χέρια μας. Και αυτή η παρουσίαση, ε, της, η ενδιάμεση παρουσίαση πριν από την ολοκλήρωση της ε, μελέτης για να μπορέσουμε και εμείς ε, να συμβάλλουμε. Αλλά επίσης πιστεύω ότι μέσα στο πλαίσιο της συζήτησής μας για την μακροπρόθεσμη προοπτική του προϋπολογισμού. Το έχουμε ήδη συζητήσει τα στοιχεία, ορισμένα από τα στοιχεία που περιέχονται στην έκθεση και ο εισηγητής επί του προϋπολογισμού ξέρει καλύτερα βεβαίως. Έχουμε πει πολλές φορές ότι χρειάζεται ένα πιο ε, ισχυρό στοιχείο ευελιξίας, ε, πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις όταν και ε, προκύπτουν και να μπορούμε να αντιδράσουμε έγκαιρα. Και αν κατάλαβα καλά από την παρουσίαση, πολλές περιφέρειες είχαν αυτή τον, τον αναγκαίο βαθμό ευελιξίας ε, ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν κονδύλια από τους προϋπολογισμούς τους να αντιμετωπίσουν καλύτερα μια μακροπρόθεσμη πολιτική προγραμματισμού. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποστήριξης των δικών μας επιχειρημάτων όσον αφορά την μακροπρόθεσμη διαχείριση του προϋπολογισμού. Και κάτι άλλο ακόμα επειδή ε, υπάρχουν πολλές περιφέρειες στην Ευρώπη και ε, καμία από αυτές δεν είναι ταυτόσιμες με μια άλλη, ε, χρειαζόμαστε μια προσαρμόσουμε πολιτική έτσι ώστε όταν θέλουμε να υλοποιήσουμε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ε, δικές τους εκάστοτε προοπτικές και βλέψεις. Μιλάμε ε, συνέχεια για την ανάπτυξη της κρίσης. Είναι προφανές ότι οι περιφέρειες διαφέρουν. Αυτό δεν χρειάζεται να ξανατονιστεί. Ευχαριστώ κύριο Σάλβες. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Καταρχάς, να συγχαρώ την ομιλήτρια για τη μελέτη. Είναι πολύ σημαντικό που ακούσαμε αυτή τη μελέτη αυτή τη στιγμή, διότι αυτά που βιώνουμε στην Ευρώπη λόγω της ε, κρίσης είναι αύξηση των ανισοτήτων και των διαφορών σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Θα ήθελα να συγχαρώ επίσης ε, τους συντάκτες της μελέτης και θα ήθελα να ρωτήσω αν είχατε δεδομένα ή κάποια προσέγγιση σχετικά με την Πορτογαλία, τη χώρα μου. Ανησυχώ πολύ για την κατάσταση λόγω της αύξησης των ανισοτήτων και των διαφορών που υπάρχουν. Σήμερα η Πορτογαλία είναι πολύ φτωχότερη, μια από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη δεδομένη στιγμή. Και μετά την κρίση όμως ο αριθμός των πλουσιών έχει αυξηθεί. Ο πλούτος τους έχει αυξηθεί κατά 9%. Σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό, που βρίσκονται στο κατόφλι της φτώχειας, αυτό έχει αυξηθεί κατά 26%. Υπάρχει τεράστια αύξηση, όχι μόνο στο χάσμα ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλουσίους, που είναι μεγαλύτερο από άλλες χώρες, αλλά και στους οικονομικούς και κοινωνικούς ε, παράγοντες που έχουν ε, ε, επιδεινωθεί. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε οποιοδήποτε στοιχείο στη μελέτη σας που επικεντρώνεται στην Πορτογαλία έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να βρούμε λύσεις για την χώρα μου. Η πολιτική συνοχής έχει συμβάλει σημαντικά, αλλά υπάρχει το θέμα της κρίσης που είναι τόσο σοβαρό που θα πρέπει να έχουμε μια σειρά από πολύπλευρες πολιτικές και κατευθυντήρες γραμμές σε οικονομικό επίπεδο, χρηματοπιστωτικό επίπεδο που είναι βασικής πρωτής σημασίας γιατί η πολιτική συνοχή από μόνη της δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιγκοέν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγητρία την εξαιρετική της μελέτη. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σχετικά με τον αντίκτυπο στην πολιτική συνοχής. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν προκύψει στο ευρωβαρόμετρο και στο, στις μελέτες του ΩΣΑ. Ε, έχουμε δει αύξηση των ανισοτήτων και της ένδυας και ο συνάδελφος είχε αναφερθεί στην Πορτογαλία. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην Ισπανία, τη δική μου πατρίδα. Όταν δούμε τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο, βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στα ευρωπαϊκά όργανα, που θεωρούνται να είναι πολύ μακριά και απομακρυσμένα από τους πολίτες. Έχουμε εκλογές στις 25 Μαΐου. Οι πολίτες αισθάνονται πολύ μακριά από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και υπάρχει ένα αίσθημα ματέωσης και απογοήτευσης γιατί κατέστη αδύνατο να υλοποιηθούν προγράμματα τα οποία ήδη είχαν εγκριθεί λόγω της απότομης πτώσης των δημοσίων δαπανών αφενός και αφετέρου της οξίας ε, πτώσης της ε, εμπιστοσύνης του κοινού στις πολιτικές συνοχής. Στην Ισπανία δεν κατορθώσαμε να δούμε ε, αυτά τα προγράμματα να έχουν κάποιο αντίκτυπο στην κρίση. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Σας ευχαριστώ και εγώ για αυτή τη μελέτη. Νομίζω είναι αξιόλογη και μας δίνει πολλά στοιχεία, τροφή για σκέψη. Ορισμένα από τα σχόλια είναι πολύ ενδιαφέροντα και καταρρίπτουν κάποιες από τις αντιλήψεις που υπάρχουν, όπως την ιδέα ότι το χάσμα βορρά-νότου, ε, δεν έχει τόση μεγάλη σημασία από τα στοιχεία και ότι υπάρχει περι, περισσότερο ε, μια διαφορά ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. Αυτό υποδεικνύει ότι θα πρέπει να είχαμε μελετήσει όλες τις χώρες. Και, άρα εγώ είμαι από την Ιρλανδία, θα ήθελα να ξέρω τις απόψεις και σχόλια σχετικά με την Ιρλανδία. Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο είναι ότι η διακύμανση έχει αυξηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εντός των χωρών έχει μείωθεί. Αυτό δεν είναι καλό συμπέρασμα για το όραμα της Ευρώπης γενικά. Είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στις πολιτικές συνοχής, όπου θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι ε, και να υπάρχει τελικά ένα ισότιμο επίπεδο, επίπεδο. Αυτή θα ήταν μια ουτοπία βέβαια αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μας ανησυχήσει αυτό. Το τελικό σημείο είναι, ε, αναφέρθηκατε σε μια σειρά από κράτη-μέλη και πώς αντιμετωπίζουν την κρίση, πώς ανακάμπτουν από την κρίση. Αλλά δεν ακούσαμε τις χώρες που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις. Ε, λοιπόν, ποιες είχαν τις καλύτερες επιδόσεις. Δηλαδή, αν ξαναρχίζαμε από το μηδέν, ποια χώρα είναι αυτή που αντιμετώπισε καλύτερα την κατάσταση και που θα μπορούσε να ήταν υπόδειγμα για τις άλλες. Αξιόλογη μελέτη, όπως είπα, αλλά χρειάζεται πολλά άλλα στοιχεία από ότι καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα την Κομισιόν αν θέλει να σχολιάσει κάποιος εκπρόσωπος. Παρακαλώ, πέστε μας ε, ποιος είστε. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ε, το όνομα μου είναι Άρτη Μπούμπιγκοκ και δουλεύω στο, στο Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης της Διεύθυνσης Οικονομικών. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε την έκτη έκθεση συνοχής η οποία θα παρουσιάσει μια πιο λεπτομερή ε, ανάλυση του τι συνέβη ε, κατά την οικονομική κρίση των ευρωπαϊκών περιφερειών. Συνεργαζόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα εν ώψη της 8ης έκθεσης ε, προόδου η οποία δημοσιεύτηκε πέρσι ε, έχουμε ήδη δημοσιεύσει ε, πολλές, αρκετά σχόλια, αρκετές παρατηρήσεις για αυτό το θέμα και αυτή η μελέτη προσθέτει ένα ακόμα ε, μια ακόμα, ε, ένα ακόμα ναι, λίθος στο οικοδόμημα της, ε, της ανάλυσης της οικονομικής κρίσης τα κατά τη διάρκεια όλων αυτών των μελετών η ανεργία έχει επιδεινωθεί, το καθάριστο, ε, τα, πολλά, τα ΑΕΠΑ καθάριστα χώρια προϊόντα έχουν επιδεινωθεί. Ε, ορισμένα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν ε, τεράστια οικονομικά προβλήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τους προπολογισμού τους. Τώρα εκτός από τις μελέτες αυτές που μας βοηθούν στις αναλύσεις, έχουμε και ε, την, ε, δημοσιο... την ε, δημοσιονομική πλευρά, την πλευρά των εισόδων του δημοσίου που όπως τονίστηκε και στη μελέτη έχουν μειωθεί και αυτό επηρεάζει άμεσα τις επενδύσεις ε, σε εθνικό επίπεδο, τις στρατηγικές επενδύσεις και επηρεάζει ιδιαίτερα την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλα τα κράτη-μέλη διότι η τοπική αυτοδιοίκηση, οι αυτοδιοικητικές περιφέρειες είναι υπεύθυνε για το 60% των επενδύσεων. Ε, υπάρχει και υπάρχουν υπάρχουν και κεντρικέ επενδύσει, παραδείγματο χάρη στον τομέα της Άμυνα. Αλλά γενικά η τοπική αυτοδίκηση, η τοπική φορή είναι υπεύθυνη για το 60% των επενδύσεων ε, στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Τι θα γινόταν λοιπόν εάν δεν είχαμε το Ταμείο Συνοχής, ε, το Περιφερειακό Ταμείο. Θα βλέπαμε ότι οι μειώσει των δημοσίων δαπανών και οι επιπτώσεις στις περιφέρειες θα ήταν πολύ μεγαλύτερες και πολύ μεγαλύτερες θα ήταν οι μειώσεις ε, και οι περικοπές των δίσεων. Είναι λοιπόν σαφές ότι οι δικές μας, τα δικά μας συμπεράσματα ε, συνάδουν με την πολιτική της ε, συνοχής. Δηλαδή η πολιτική συνοχής η βοηθάει την επίλυση των προβλημάτων, τη διαφορετική αναδιάρθρωση, την ενίσχυση του, κεφα, του κεφαλουχικού δυναμικού των, των περιφερειών, την εφαρμογή ευέλικτων πολιτικών κλπ. Ε, πρέπει λοιπόν να ε, αναγνωρίσουμε την βοήθεια του, της πολιτικής συνοχής, να υλοποιήσουμε διορθωτικές ε, μεταρρυθμίσεις, αλλά επίσης να υποβοηθήσουμε με συγχρηματοδότηση τις επενδύσεις. Και σε πολλές χώρες τα διαφορετικά ταμεία έχουν βοηθήσει σημαντικά ε, τις επενδύσεις. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμεσα την έκτη έκθεση συνοχής και θα τη δημοσιεύσω σύντομα όπου θα δείτε τα συμπεράσματά μας σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαν Ρόι, παρακαλώ να λάβει το λόγο και μετά θα απαντήσει η δόκτωρ Μίλιο. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου αναφέρεται στο εξή σημείο. Ζητήσαμε να γίνουν αλλαγές στην πολιτική, δεν υπάρχει αμφιβολία, διότι είδαμε σαφώς ότι έχουν μειωθεί, έχει μειωθεί η συμβολή κρατών μελών που αντιμετωπίζουν σοβαρότατες οικονομικές κρίσεις. Ζητήσαμε λοιπόν αλλαγές στους κανονισμούς, στους συναφείς κανονισμούς. Έχετε μελετήσει λοιπόν αυτό το θέμα της μείωσης των, των ιδίων πόρων. Επίσης, επιπτώσεις ε, και χρηματοδοτήσεις από τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία. Έχετε δει πώς έχει διακυμανθεί η ενίσχυση, οι χρηματοδοτήσεις μεταξύ φτωχότερων και πλουσιότερων περιοχών μελετήσατε πώς τα κοινωνικά ταμεία ε, μπόρεσαν να έχουν κάποια επίπτωση αντιμετώπισης ή πρόεδρος. <coughs> Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει ζητήσει το λόγο. Η κυρία Μίλιο θα πάρει το λόγο. Στον πρώτο κύριο που έθεσε ερωτήσεις αναγνωρίζω τη σημασία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάκαμψης. Δεν ήταν βασικό θέμα μας το πώς εφαρμόστηκε, δεν ήταν αυτό το αντικείμενο αν θέλετε. Εμείς ερευνήσαμε τις επιπτώσεις της κρίσης στα κράτη-μέλη και πώς η περιφερειακή πολιτική ανταποκρίθηκε. Οπότε στην ουσία η νέα ερώτηση την οποία θέτεται είναι πολύ ε, ευρία και πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό το οποίο μπορώ να πω αν μου επιτρέπετε είναι ότι για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης αυτό το οποίο είδαμε, αυτό το οποίο μελετήσαμε είναι το τμήμα του προγράμματος αυτού που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι δυνατότητες ε, σωστότερης χρήσης ε, και απορροφητικότητας ε, των διαθεσίμων πιστώσεων. Αυτό ήταν το βασικό χαρακτηριστικό. Ξέρω ότι ασχολείται το πρόγραμμα αυτό κυρίως με θέματα ενέργειας και υποδομών, αλλά δεν ήταν το αντικείμενο της μελέτης μας. Αν πάτε στην διαφάνεια 27 θα δείτε ότι κάνω μία συγκεκριμένη παρατήρηση ότι η Ιταλία είναι μία χώρα στις οποίες δυστυχώς η προσθετικότητα μειώθηκε και ε, τα κοινοτικά ποσά ήταν ε, τα αποκλειστικά μέσα μερικές φορές για ορισμένου τομείς. Δεν μπορώ ε, από τα 25 λεφτά που είχα στη διάθεσή μου να σταθώ περισσότερο στα της ε, προσθετικότητας, αλλά όπως είδατε αναφέρθηκα σε αυτό. hard outcomes και soft outcomes. Τι είναι αυτά. Αυτά είναι ε, στην ουσία παρατηρήσεις κλείνοντας. Εγώ είμαι πανεπιστημιακός και στην ουσία ε, βλέπω ποια είναι τα όρια κάθε φορά της προσπάθειας την οποία κάνουμε. Συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στα hard outcomes. Τι εννοούμε. ΑΕΠ, ανάπτυξη του ΑΕΠ, ποσοστά απασχόλησης, ποσοστά ανεργίας. Όταν μιλάμε σαν παράδειγμα για απασχόληση, αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε hard outcome. Προσπαθούμε να δούμε το τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί στην απασχόληση στήριξη στους πολίτες να αποκτήσουν ικανότητες, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους, να μειώσουν τον χρόνο μετακίνησης προς την εργασία. Όλα αυτά επηρεάζουν την απασχόληση. Ε, όταν βλέπουμε τα ποσοστά μερικές φορές αγνοούμε το τι οδήγησε στα ποσοστά αυτά ανεργίας ή απασχόλησης. Εμείς λοιπόν βλέπουμε ότι πρέπει να κάνουμε μια ισχυρή ποσοτική ανάλυση την οποία θα πρέπει να συνδυάσουμε ε, με μεγαλύτερες ποιοτικές εκλεπτύνσεις αν θέλετε στη σκέψη μας και στα σχόλιά μας. Για τη δεύτερη ερώτηση αναφερθήκατε στην ευελιξία. Νομίζω ότι η ευελιξία έχει βοηθήσει πάρα πολύ τις διάφορες περιφέρειες, αλλά όπως είπα και στην καταληκτική διαφάνεια είναι ε, εξαιρετική η ευελιξία, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να υπονομεύει τον έλεγχο. Αν ευελιξία σημαίνει συνεχής αλλαγή κανόνων, μπορεί να επηρεάσει την διαφάνεια αρνητικά, την αλλαγή των κανόνων, γιατί αλλάζουν οι κανόνες κτλ. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία λοιπόν ανάμεσα στην δυνατότητα ελέγχου και ε, την ευελιξία. Χαίρομαι που βρήκατε για τα συμπεράσματα στον τομέα της πολιτικής συνοχής για την γεωγραφική διαφοροποίηση ενδιαφέροντα. Το θέμα δεν είναι να διαφοροποιούμε ανάμεσα στις περιοχές σύγκλησης και τις περιοχές ανταγωνιστικότητας. Αλλά και στο εσωτερικό των περιφερειών σύγκλησης κάποιες περιοχές είναι ισχυρότερες από άλλες. Το ίδιο φάνηκε και στην Πολωνία. Κάποιες χώρες συνοχής, συγκλήσης, συγγνώμη, είναι ισχυρότερες από άλλες. Κάποιες περιοχές στο εσωτερικό μιας χώρας είναι ισχυρότερες από άλλες. Παίζει ρόλο λοιπόν η διαφοροποίηση αυτή στην ερώτηση για την Πορτογαλία και για τα δεδομένα για την Πορτογαλία. Η ποσοτική ανάλυση όπως είπα, η μελέτη διαιρείται σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι ποιοτικό και το δεύτερο ποσοτικό ή αντίστροφα. Σε επίπεδο ποσοτικό εμείς συλλέξαμε στοιχεία από το σύνολο των κρατών μελών και <clears throat> χρησιμοποιήσαμε 28 δίκτες για κάθε περιφέρεια. Εγώ δεν θα ήθελα να παρουσιάσω στην παρούσα φάση, αλλά όταν δημοσιευθεί πλήρως η μελέτη θα υπάρξουν τα επιμέρους αυτά στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει. Τα υπόλοιπα σχόλια ήταν σχόλια συμφωνίας με τα συμπεράσματα. Είμαι στη διάθεσή σας να συνεχίσω την επικοινωνία μαζί σας και να συζητήσω αν πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει θετικά στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής. Ξέρετε ότι η περιφερειακή πολιτική χρησιμοποιήθηκε για να αναπληρώσει την κατάρρευση ουσιαστικά πολλών τομέων και πολλών μορφών, διαφορετικών μορφών χρηματοδότησης. Τώρα για το κοινωνικό ταμείο, τελευταία ερώτηση. Η μελέτη αυτή αφορά τα θέματα συνοχής περισσότερο. Βέβαια εξετάσαμε και τα κοινωνικά και είδαμε τις επιπτώσεις της εφαρμογής των κοινωνικών, της παρέμβασης των κοινωνικών ταμείων. Ιδιαίτερα στον τομέα της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της κρίσης του κοινωνικού ταμείου ε, καταπολεμήθηκε η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Βασικό, ε, βασική συνέπεια της κρίσης. Thank you very much also for your... Ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρος. Σας ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση. Ήταν μια διάμεση φάση αυτή. Ακόμα δεν έχουμε ολοκληρωμένη τη μελέτη στα χέρια μας. Εάν η μελέτη αυτή διάτεθεί πριν από τις ε, ευρωεκλογέ, είμαι βέβαιη ότι πολλοί συνάδελφοι θα ήθελαν να την ε, μελετήσουν, να τη διαβάσουν, αλλά ε, σίγουρα θα επανέλθει το θέμα στην επόμενη θητεία και στις επόμενες συνεδριάσεις του νέου σώματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ευχαριστούμε την κυρία Μίλιο για την συμβολή της στην συζήτησή μας. Ε, και τώρα ε, μπορούμε να ήδη βλέπω τους ομιλητές του επόμενου θέματος. Δεν ξέρω αν όλοι είναι εδώ. Ε, ορισμένοι ακόμα προσέρχονται στην αίθουσα. Μπορούμε να αρχίσουμε γιατί η πρώτη ομιλήτρια επί του θέματος είναι εδώ. Το θέμα μας είναι μικροχρηματοδότηση και πολιτική συνοχής και όσοι έχετε συμμετάσχει στις συζητήσεις αυτές στο Κοινοβούλιο ε, συζήτηση για την έξοδο από την κρίση πολλοί συνάδελφοι έχουν πει ότι ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σε χρηματοδότηση, σε πιστώσεις και γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το όλο θέμα της μικροχρηματοδότησης, microfinance και πώς μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στην Ευρώπη. Έχουμε τρεις ομιλητές και θα αρχίσουμε με την κυρία Ιζαμπέλ Ντεσρέβερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο η οποία είναι υπεύθυνη στρατηγικό προγραμμάτων. συνεχεία ακούσουμε τον κύριο Έριξον ε, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την κυρία Μαρία Νόβακ που είναι πρόεδρος της ε, AD International. Νομίζω ότι όλοι είναι εδώ και δίνω το λόγο στην κυρία Ντεσρίβερ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε σε αυτή τη συνεδρίαση σήμερα το πρωί. Είναι μεγάλη τιμή μου που θα μοιραστώ μαζί σας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης Jasmine στην πιλωτική φάση που ξεκίνησε από εσά, κυρία Χιούπνερ, το 2008. Όλα ξεκίνησαν με μια ανακοίνωση από την Κομισιόν το 2007 για την μη μικρο, τις μικροπιστώσεις ως τρόπος στήριξης της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με βάση αυτή την ανακοίνωση αναπτύχθηκε το η πιλωτική φάση του Jasmine με δύο άξονες. Ο πρώτον, η τεχνική βοήθεια σε επιλεγμένους δικαιούχους. Δικαιούχους που είχαν επιλεγεί ε, μετά από προκήρυξη ε, ενδιαφέροντος και δεύτερος, δεύτερος άξονος ε, σε ολόκληρο τον ε, τομέα, σε ολόκληρο τον κλάδο για ε, θέματα μικροπιστώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας ο, Καλής Πρακτικής για την ε, παροχή μικρό χρηματοδότησης δεν ήταν μέρος της αξιολόγησής μας, αλλά θα ήθελα να πω μερικά λόγια για αυτό το έγγραφο. Είναι ένα έγγραφο που είναι ένας οδηγός, ο οποίος καθίσταται όλο ένα και πιο σημαντικός στον κλάδο μας. και αποτελεί τώρα και πυλώνα της τεχνικής βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κώδικας ορθής πρακτικής είναι μία σειρά από πρότυπα. Είναι μια, ένας κατάλογος ε, από ρήτερες. είναι αυτό το έγγραφο που βλέπετε εδώ, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον κλάδο τον τομέα και μας βοήθησε να δούμε ποιες είναι οι σημαντικές ρήτρε έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους παρόχους μικροχρηματοδότησης να βελτιώσουν ποιότητα της, δουλειά τους, της δουλειάς τους, να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια ε, στον τομέα της, ε, των εκθέσεων κλπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους παρόχους μικροπιστώσεων, μικροχρηματοδότησης, διότι δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι. πόροι με Και αυτή τη στιγμή οι επενδυτές ε, είναι πιο επιλεκτικοί στους παρόχους μικροχρηματοδότησης. Γι' αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο αυτό. Ακούω από μικρούς οργανισμούς που λένε ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό το έγγραφο, διότι μας βοηθάει να δούμε ποια είναι τα σημαντικά κριτήρια και στοιχεία για να ε, κάνουμε την επιλογή μας. Από το 2013 έχουμε και την μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί με τη στήριξη του Πανεπιστημίου του Σάλφορτ, έτσι ώστε να μπορούμε να αναλύουμε αν οι ρήτρε του κώδικα εφαρμόζονται καλά από κάποιον οργανισμό ή όχι. Επίσης αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση από τους αξιολογητές για να επαληθεύσουν την ορθή υλοποίηση του κώδικα. Θα συνοδεύεται και από το Jasmine Online που είναι μια ασφαλής ε, εφαρμογή στο διαδίκτυο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι πάροχοι για... και αυτά συνιστώνται από τον κώδικα ορθής πρακτικής. Τώρα να επανέλθω στην αξιολόγησή μας. Η στόχη της αξιολόγησης ε, της πιλωτικής φάσης Jasmine ήταν να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα. Ποια είναι τα διδάγματα που έχουμε αποκομίσει, ποιες είναι οι συστάσεις το πεδίο εφαρμογή από το 2008 μέχρι το 2012. Γνωρίζοντας ότι οι πρώτοι δικαιούχοι έλαβαν τη στήριξη του Jasmine το 2011, διότι πήρε χρόνο η όλη η θέσπιση και η προκήρυξη κλπ. Αναλύσαμε ε, τη στήριξη που ε, περιεχόταν στον κλάδο και έγινε η επιλογή των δικαιώχων. Εδώ βλέπουμε κάποια από τα ευρήματα από την αξιολόγηση αυτή που έγινε από το ICFTHK. Αυτό που συνοψίζει καλύτερα τα ευρήματα είναι ότι το Jasmine βοήθησε να καταστήσουμε τον τομέα μικροχρηματοδότησης πιο επαγγελματικό. Δηλαδή, η παρόχη μικροχρηματοδοτήσεων ε, μας είπαν ότι τους βοήθησε να βελτιώσουν τη λειτουργική τους ικανότητα, την παραγωγικότητα, αλλά και τις εξωτερικές σχέσεις τους μέσα από τα εργαστήρια, διότι όλοι είναι μέλη δικτύων, αλλά και τα εργαστήρια τους βοήθησαν να ε, κάνουν επαφές και να, να τους ε, εκτιμήσουν καλύτερα οι πελάτες τους, διότι αξιοποίησαν αυτή την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Επίσης, ε, αναπτύχθηκε η προώθηση των ε, ιδεών και των αντιλήψεων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Μας είπαν επίσης ότι τους έδωσε πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης τα οποία δεν θα μπορούσαν να καλύψουν από μόνοι τους. Άρα υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση. Τώρα, Ποιες είναι οι συστάσεις που λάβαμε. Υπάρχει ένα αίτημα για ευρύτερη κατάρτιση, πιο πολύ κατάρτιση. Κάποιοι θα ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα προγράμματα κατάρτισης και ε, να μην σχετίζονται απαραίτητα με το Jasmine. Επίσης, μια άλλη σύσταση, να υπάρχει ένα πιο αναπτυγμένο μέτρο του κοινωνικού αντίκτυπου, να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα. Αυτό μπορεί να επεκταθεί μέσω του Jasmine Online. Η φόρμουλα των εργαστηρίων επίσης ε, υπήρχε μια σύσταση όπως ε, να υπάρχουν πιο, ε, πιο δυναμικά εργαστήρια με μεγαλύτερη συμμετοχή. η εναρμόνιση επίσης των ε, εκθέσεων των ε, οργανισμών ε, διαπίστευσης της χρηματοπιστωτικής ικανότητας. Σε άλλες φορές θα συμβάλλουν κάπως στην υπηρεσία αυτή, ενώ μέχρι τώρα ήταν δωρεάν. Το τι θα κάνουμε τώρα, ποια συνέχεια θα δοθεί θα συνεχιστεί η τεχνική βοήθεια και στην ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων στη βοήθεια των παρόχων μικροπιστώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τους επενδυτές, τους ενδυνάμει επενδυτές, όπως είπα και πριν, αλλά και αυτούς τους οργανισμούς μικροχρηματοδότησης, που είναι ένα σύνδεσμος με τους πελάτες τους, με τις εταιρείες μικροχρηματοδότησης, μικροπιστώσεων, έτσι ώστε η πάροχοι μικροπιστώσεων είναι ο άμεσος σύνδεσμος και είναι σημαντικό να παρέχουν ποιοτική στήριξη. Είναι αυτό το οποίο κάνουν ήδη και αυτό τους κάνει να, διαφέρει, να διαφέρουν από τις τράπεζες. Οι πάροχοι μικροπιστώσεων έχουν και αυτό το κοινωνικό στοιχείο. Είναι ένα χέρι βοηθείας που παρέχουν. Παρέχουν στήριξη, βλέπουν τα προγράμματα και τα έργα μαζί με τους πελάτες τους και ε, πρέπει και αυτοί όμως να τύχουν στήριξης. Γιατί όπως είπα βοηθάνε τους οργανισμούς μικροπιστώσεων και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί οι οργανισμοί είναι περίπου το 50% ε, των θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, είναι σημαντικό να παρέχουμε στήριξη σε αυτούς και ναι, η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη. Συνεργαζόμαστε με την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και την Γενική Διεύθυνση για τις Περιφέρειες και η DG Regio αυτή τη στιγμή αναπτύσσει την πλατφόρμα τεχνικής βοήθειας που είναι ένα πλαίσιο όπου η τεχνική βοήθεια θα αναπτυχθεί εντός της ε, Κομισιόν όπου διαφορετικές γενικές διευθύνσεις θα συμμετέχουν και εκεί ε, θα συμπεριληφθεί και η τεχνική βοήθεια προς τους παρόχους μικροπιστώσεων. Αυτό που θέλουμε επίσης να αναπτύξουμε περαιτέρω και ο συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, Ταμείο Επενδύσεων, με ε, συγχωρείτε, είναι να ε, έχουμε τεχνική βοήθεια και το EPMF, γιατί υπάρχει σύνδεσμος ανάμεσα στα δύο. Τώρα, Ας δώσουμε το λόγο στον κύριο Έριξον, ο οποίος θα σας αναλύσει το EPMF. Ευχαριστώ κύριε Αντεσίδερο, κύριο Πέρα Έριξον. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσω για την μικροχρηματοδότηση. Ξεκίνησε το 11, η νομική βάση είναι τον Απρίλιο του 10. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και διαχειριστής είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων προβλέπεται ένα συγκεκριμένο ποσό για τα μέσα χρηματοδότησης, 23 εκατομμύρια για τα μέσα εγγυήσεων, η μόχλευση είναι 5, 100 δηλαδή εκατομμύρια από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία θα διαθέσουν 500 εκατομμύρια μικροπιστώσεων. Υπάρχουν στόχοι κοινωνικής συμπερίληψης, και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Καλύψαμε 18 χώρες μέχρι τώρα. Το επόμενο τρίμηνο θα καλύψουμε άλλες δύο, θα φτάσουμε λοιπόν τις 20 χώρες. Είμαστε επίσης και με κάποιες άλλες χώρες σε διάλογο. Ένας από τους λόγους που δεν έχουμε 28 χώρες ε, είναι ότι εμείς προσπαθούμε να συμπληρώσουμε τα εθνικά συστήματα μικροχρηματοδότησης είτε από ε, ιδιωτικούς πόρους είτε από το δημόσιο της κάθε χώρας. Θα φτάσουμε τα 200 εκατομμύρια σε αυτό το τρίμηνο, 40% έχουμε διαθέσει δηλαδή, πάμε καλά. Νομίζω ότι έχουμε μια κοινωνική εισχώρηση πάρα πολύ ικανοποιητική και έχουμε φτάσει σε ποσοστά απορρόφησης ανά περίοδο στο 97%. Κυρίως δίνουμε κάποιες ε, δυνατότητες εγγύησης δανείων. Το μέσο εγγυήσεων χρησιμοποιείται πλήρως και χρησιμοποίησαμε επίσης και τα δύο τρίτα των διαθέσιμων ταμείων για τα μέσα χρηματοδότησης. Αυτό εδώ δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε. Η κόκκινη γραμμή δείχνει το πού βρισκόμαστε τώρα στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2013. Βλέπουμε ότι στο τέλος του 2017 θα έχουμε ξεπεράσει τον στόχο των 500 εκατομμυρίων που ήταν ο αρχικός στόχος. Το ίδιο γράφημα δείχνει ότι έχουμε δείχνει και τον αριθμό των δανείων και όχι τόσο το ύψος, το συνολικό, μέχρι το 2017 θα έχουμε επιτρέψει να διατεθούν 46.000 δανειακές διευκολύνσεις. Στον τομέα της κοινωνικής εισχώρησης, στους μικροδανειολήπτες δηλαδή, εδώ βασίζεται σε 12.000 περίπου το στατιστικό δείγμα και βλέπουμε ότι έχουμε ειδικέ αναφορές επιτυχίας για το 97%. Το 63% είναι άνδρες, 37 γυναίκες. Όταν μιλάμε για μικρό δανειοδοτήσεις βλέπουμε ότι έχουμε κάποια επιμέρους στοιχεία και η εισχώρηση στον στόχο των ανέργων πάνω από το 50% αυτών που πήραν τα δάνεια δεν ήταν δραστηριοποιημένοι επαγγελματικά ή ήταν απλά άνεργοι. Σε σχέση με τη δημιουργία των θέσεων απασχόλησης μέχρι τώρα έχουμε κάποια προκαταρκτικά στοιχεία σε κάποιες περιπτώσεις ε, έχουμε πολύ ικανοποιητικές, ε, ικανοποιητικά παραδείγματα όπως ε, πάνω από ένα εκατομμύριο στην Πολωνία. σε σχέση με τις ομάδες στόχους. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι αποφελήθηκαν είναι αυτό που ονομάζουμε startups, μικρομεσαίες που ξεκινούν και δεν είναι πάνω από 2-3 ετών το 44% δεν υπάρχουν ούτε καν ένα χρόνο πριν. Έχουμε συγκεντρώσει την προσοχή μας λοιπόν η ενδιάμεση σε 100% εταιρείες οι οποίες ξεκινούν τώρα. Σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης βλέπουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις Βλέπουμε ότι στη Βουλγαρία σαν παραδείγμα το 1 τρίτο αυτών που πήραν τα χρήματα ήταν της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή δεν είχαν καμία εκπαίδευση. Έχουμε επίσης μια καλή εισχώρηση στη μειονότητα των Ρωμά στη Βουλγαρία και βλέπουμε ότι με το BCP στην Πορτογαλία το 90% αυτών που πήραν χρήματα είναι από την δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με, κοινωνική, με τους δείκτες κοινωνικής εισχώρησης. Να πω ότι στηρίζουμε τους νέους επιχειρηματίες σε ηλικιακό επίπεδο. Κάτω από 25 ετών είναι το 6%. Έχουμε κάποιους ενδιαμέσους σε διάφορες χώρες όπου πάνω από το 20% ανήκουν στην κατηγορία κάτω των 25 ετών. Αν δείτε επίσης τις ομάδες στόχων, το 2% έχουν δηλώσει ότι ανήκουν σε μειονότητες. Αυτό είναι βέβαια μια δυνατότητα αυτοδήλωσης, οπότε υπάρχουν πολλά στοιχεία που δεν έχουμε εδώ πέραν από αυτούς τους στόχους σε ενδιάμεσο επίπεδο βλέπουμε ότι οι κάποιοι ενδιάμεσοι έχουν ιδιαίτερα καλή σχέση με τις μειονότητες όπως το Patria Credit, το Sverbank Slovenia και το Microfond. Τώρα το Jasmine TA, συμπληρωματικότητα με το Jasmine TA. 70 έχουν επωφεληθεί από αυτή την ιστορία, 12 έχουν εποφεληθεί είτε μέσω εγγυήσεων είτε μέσω άμυσης χρηματοδότησης, ε, κάποιοι έχουν παραπεμφθεί για αποκλειστική χρηματοδότηση από το Just Mean TA. και το 30% από το Jasmine TA προσπαθούν να υποφεληθούν επίσης και από τις δυνατότητες χρηματοδότησης τις υπόλοιπες. Σε κάποιους τομείς έχουν υπάρξει βελτιώσεις. Προγράμματα δηλαδή για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία. Ενισχύουμε επίσης ε, τη δράση των μη πιστοτικών, μη τραπεζικών πιστοτικών ιδρυμάτων. Και βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα και σε επίπεδο καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και σε επίπεδο κοινωνικής εισχώρησης είναι πολύ καλύτερα από ό,τι οι παραδοσιακές τράπεζες. Ξέραμε ότι η αγορά αυτή ήταν ιδιαίτερα ετερογενής, σε πάση περιπτώσει, και είδαμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά προγράμματα προσφερόμενα και γι' αυτό επιλέξαμε κάποια προγράμματα όπως οικονομική στήριξη, όπως επίσης ε, ε, οι εγγυήσει ή οι άμεσες χρηματοδοτήσεις. Χρειάστηκε να προσαρμόσουμε λοιπόν τις δυνατότητες τις οποίες ε, είχαμε μέχρι τώρα βέβαια υπάρχουν κάποιοι νομικοί περιορισμοί εδώ, σαν παράδειγμα δεν μπορούν οι εταιρείε αυτές να εκδώσουν μετοχές κτλ. Θα ζητήσω τώρα από την κυρία Νόβακ να πάρει το λόγο και να αναφερθεί λίγο και στο όργανο το οποίο εκπροσωπεί η κυρία Νόβακ. Ευχαριστώ.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 σε αυτό το θέμα. Εγώ δεν θα μιλήσω για τα μέσα, για τα διάφορα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά θα μιλήσω περισσότερο από την πλευρά της πολιτικής συνοχής που πιστεύω είναι πολύ σημαντική για τη μικροχρηματοδότηση. Καταρχάς, η ανάπτυξη του όλου θέματος της μικροχρηματοδότησης ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις μελλοντικές της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και πολιτικής συνοχής. 92% όλων των επιχειρήσεων ε, στην Ευρώπη είναι μικροεπιχειρήσεις με λιγότερο από 50 απασχολούμενους και υπάρχει επίσης και ένας ανεπίσημος άτυπος τομέας ε, που δεν ξέρουμε ακριβώς τα αριθμητικά δεδομένα αλλά αντιπροσωπεύει περίπου το 10 με 15% του ΑΕΠ. Βλέπετε λοιπόν και ο τελευταίος δείκτης είναι ο ενεργός πλησισμός κάτω από το όριο φτώχειας 28 εκατομμύρια άτομα. Αν εξετάσουμε τώρα τις μελλοντικές προοπτικές, είναι σημαντικό να πούμε ότι διαγράφονται πολύ σημαντικές τάσεις οι οποίες βασίζονται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών, στην μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους που συμβαίνει βέβαια και αυτή η εξέλιξη μας οδηγεί περισσότερο στην ανάγκη ανάπτυξης μικρών παραγωγικών μονάδων ε, οπότε προφανώς το μέσο της μικροχρηματοδότησης γίνεται ένα σημαντικό μέσο, ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη. Θα ήθελα να σας δείξω δύο ε, γραφήματα ε, ε, των πίνακα αυτών που δείχνει μία εξέλιξη συγκριτική του τομέα των υπηρεσιών και της απασχόλησης στον τομέα αυτών. Το πράσινο είναι ακριβώς η απασχόληση στο, στο τρίμηνο και η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει την βιομηχανία και την κατασκευή. Η πράσινη γραμμή είναι το μέσο των υπηρεσιών. Βλέπετε λοιπόν ε, και αφορά, αφορούν τα, το, το γράφημα αυτό, πίνακα σε αυτό αφορά τη Γαλλία και βλέπετε ίσως σε άλλες χώρες να υπάρχει μια διαφορετική διακύμαση, αλλά βλέπετε ακριβώς πόσο αναπτύσσεται ο τριτογενής ε, τομέας και πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει λοιπόν για μικροχρηματοδότηση αυτού του τομέα. Η Ιζαμπέλ ανέφερε αυτή την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της χρηματοδότησης ως εργαλείο μέσων μέσον στήριξης της, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Και ακόμα ισχύει αυτός ο στόχος, σαφώς. Ε, είχα τότε συνεργαστεί στην προετοιμασία αυτής της ε, μελέτης μαζί με τον κύριο Φιλίπ Ντελβό, ο οποίος ήταν ο προκάτοχος της θέσης της κυρίας Σρίβερ, ε, και με τον προκάτοχο της, ε, του κυρίου Έριξον και ε, αυτές οι τάσεις τότε είχαν βασιστεί σε λανθασμένες τάσεις διότι μην ξεχνάτε ότι τότε είχαμε πρωτοαρχίσει τη συζήτηση για την μικροχρηματοδότηση και είχαμε πει τότε ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι νομικές και ε, θεσμικές ε, υποδομές, όλο το περιβάλλον το θεσμικό και το νομικό στα κράτη-μέλη. Και από τότε που τα είπαμε αυτά, το μόνο που έχει γίνει είναι μία ε, διάσκεψη η οποία οργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου του 2011. Αυτά όλα τα είχαμε πει το 2007. Είχαν υποθεί μάλλον το 2007 από τους προκατόχους. Και οργανώθηκε αυτή η διάσκεψη η οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δεν επακολούθησε κάποια ε, ε, ενθάρρυνση για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και καλά αλλά θα έπρεπε να, είχαν, να είχε προσφερθεί μια πρακτική υποστήριξη για την αλλαγή μεταρρύθμιση αυτού του νομικού και θεσμικού πλαισίου. Η δεύτερη τάση τότε, την οποία είχαν καταλήξει, ήταν πρέπει να αλλάξει περαιτέρω όλο το επιχειρησιακό ε, περιβάλλον προς όφελος ε, του επιχειρησιακού πνεύματος. Ας μην ξεχνάμε ότι όλο το νομικό πλαίσιο της εργασίας τότε ε, είχε προσαρμοστεί περισσότερο στις ανάγκες μεγάλων επιχειρήσεων. Ε, φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ε, ανομαλία στην, στην εμφάνιση των διαφανειών στον πίνακα και κάτι δεν πάει καλά στην σειρά της εμφάνισης των διαφανειών της ομιλήτρια. Ε, λοιπόν, ε, το νομικό πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, τότε ήταν περισσότερο ε, προσανατολισμένο προς τις μεγάλες επιχειρήσεις και δεν είχε προσαρμοστεί τότε στους αυτοαπασχολούμενους ή στις ανάγκες για μικροχρηματοδότηση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Γαλλία Είχαμε τότε, περάσει, είχε περάσει ένας νόμος για τους αυτοαπασχολούμενους που είχε απλοποιήσει το σύστημα και επέτρεπε στα άτομα αυτά να πληρώσουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, όχι πριν, προκαταβολικά πριν εισπράξουν ε, λεφτά, αλλά μετά και σε τρία χρόνια ένα εκατομμύριο νέες μικροεπιχειρήσεις καταχωρήθηκαν στο Μητρό. Οπότε βλέπετε ότι μια τέτοια αλλαγή είχε τεράστια επίπτωση και μια τέτοια βελτίωση του νομικού πλαισίου είχε μια τεράστια βελτίωση στο επιχειρηματικό τομέα και πιστεύω ότι αυτό ε, θα μπορούσε να το ενισχύσει αυτή την εξέλιξη και τον προσανατολισμό θα μπορούσε να βοηθήσει και η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τρίτη τάση είναι η προώθηση ε, της διασποράς των βέλτιστων ε, πρακτικών. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι πέραν της ε, δημιουργίας δυναμικού του capacity building υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα στην πρόσβαση. Παραδείγματο χάρη στο να διευκολύνουμε την πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα διαστροτικά ταμεία. Πρόσβαση των επιχειρήσεων. Πρόσβαση των επιχειρηματιών. Επίσης, ε, όσον αφορά τις ε, υποστηρικτικές εργασίες τις οποίες δεν μπορούν να κάνουν οι μικροεπιχειρήσεις αν δεν έχουν την ε, μικροπιστώση, τη βοήθεια δηλαδή από το πλαίσιο αυτό. Η τέταρτη τάση ήταν η προσφορά, η παροχή συμπληρωματικών κεφαλαίων από μικροχρηματοδότης, τραπεζική και μη τραπεζική. Εδώ είχαμε εξετάσει τα διασωτικά ταμεία και την πρόοδο αυτής της, ε, του εργαλείου, αυτού του μέσου. Και είναι πολύ σημαντικό να καταγράψουμε τι έχει γίνει. Όμως, παρόλες τις κατά μέρος επιτυχίες, βλέπουμε ότι δεν προσαρμόζεται πάντοτε το πρόγραμμα αυτό στην πραγματικότητα των ε, ιδρυμάτων των φορέων μικροχρηματοδότησης. Παραδείγματος χάρη, πάνω από το ίμιση των μικροπιστωτικών ιδρυμάτων έχουν διαθέσει λιγότερο από 100 πιστώσεις, 100 δάνεια το χρόνο. Έχουν δανειοδοτήσει δηλαδή λιγότερο από 100 φορές το χρόνο, το οποίο δεν είναι και πολύ χρήσιμο όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να ή να βελτιωθούν ή να σταματήσουν τη λειτουργία τους εφόσον είναι αναποτελεσματική. Πιστεύω ότι ε, από τη φύση του το σύστημα δεν είναι προσαρμοσμένο σε αυτόν τον τύπο των προβλημάτων, διότι στα ε, ε, ε, χρηματοδοτικά ιδρύματα είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στην ενίσχυση των κεφαλαίων, στην κάλυψη υψηλού κόστους μεγάλων επιχειρήσεων και το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι ότι η, η μικροχρηματοδότηση των νέων επιχειρήσεων που ξεκινούν έχουν τεράστιες δυσκολίες πρόσβασης σε αυτό το μέσον, σε αυτές τις πιστώσεις. Καταλήγοντας λοιπόν θέλω να πω ότι η μικροχρηματοδότηση είναι ένα μέσον το οποίο πρέπει να προσανατολίζεται και να βασίζεται στην πραγματική οικονομία, στα πραγματικά στοιχεία. Μπορεί να γίνει ένα βασικό εργαλείο της πολιτικής συνοχής, διότι προσανατολίζεται σε άτομα, σε επιχειρηματίες ε, που ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Στοχεύει στην απασχόληση των νέων, δεν ε, στοχεύει μόνο στην οικονομική ενσωμάτωση, υποστήριξη, αλλά και στην περιφερειακή ενσωμάτωση και πιστεύω ότι μπορούν να αναπτυχθούν τα μέσα αυτά με, με πολύ σημαντικό τρόπο για να ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα και να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες. Βλέπετε ότι από το 2010 το πρόγραμμα προόδου της μικροχρηματοδότησης έχει υποστηρίξει 9.000 μικροεπιχειρηματίες με 80 εκατομμύρια ευρώ. Ε, και ο ανεργός πληθυσμός, όπως είπαμε, κάτω από το όριο της φτώχειας είναι 28 εκατομμύρια. Βεβαίως είναι μία μικρή σοδιά αυτή, ένα περιορισμένο αποτέλεσμα αν θέλετε, αλλά έχουμε ένα τεράστιο περιθώριο προόδου για την ανάπτυξη αυτής ε, της απασχόλησης και αυτού του είδους ε, των πιστώσεων. Μεγάλο, μεγάλες προοπτικές δηλαδή και ταυτόχρονα ε, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη συνοχή οικονομική και περιφερειακή. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, τα πάντα να τα αναμένουμε, ε, να τα κάνει η Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους ενθαρρύνουμε, να ασκήσουμε πίεση δράσεις, αλλά πρέπει να παρουσιάσουμε σωστά ε, το δυναμικό αυτής της ε, μικροχρηματοδότησης, γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν τη σημασία που, έχει αυτό το μέσον ε, μικροχρηματοδότησης από μη τραπεζικές πηγές. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη του κοινού μας στόχου της δημιουργίας ευημερίας. Σας ευχαριστώ. Η Κωνσταντσε Κρέλ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ για τις, ε, τις ε, εισηγήσεις σας και των τριών ομιλητών. Η παροχή μικρών μικροδανείων είναι ένα πάρα πολύ σον μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Και μετά από τις εισηγήσεις που άκουσα έχω δύο ερωτήσεις. Θα με ενδιέφερε εάν έχετε εμπειρία, αν ξέρετε, εάν υπάρχουν και τι ποσοστά λάθους φαλμάτων υπάρχουν μέσα σε αυτό το σύστημα μικροχρηματοδότησης. Μάλλον απαντήθηκε το ερώτημά μου από την τελευταία παρέμβαση το ότι σχετικά μικρό το περιθώριο. Και δεύτερον θα ήθελα να ξέρω ότι πόσο μεγάλη είναι ανάγκη ε, αυτού του τομέα. Δηλαδή, πέραν από τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάσατε για το τι έχει υλοποιηθεί, τι είδους ανάγκες υπάρχουν ακόμα. Και η τελευταία παρέμβαση μας έδειξε σαφώς ότι πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν πρόσβαση ακόμα σε αυτό το μέσον. Ρωτώ λοιπόν, δεδομένου ότι θα έχετε μελετήσει τους νέους κανονισμούς για τη νέα πολιτική, μελλοντική πολιτική συνοχής, πιστεύετε ότι αυτοί οι νέοι κανονισμοί θα παρουσιάσουν καλύτερες δυνατότητες, θα βελτιώσουν την κατάσταση ή θα συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει. Η Πρόεδρος, για, για να μπορώ και εγώ να συμπληρώσω αυτά που είπε η Κωνσταντσα, όταν διαπραγματευόμεσα τα ε, δημοσιονομικά εργαλεία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο της συνοχής, είχαμε πει ότι τα ε, χρηματοδοτικά εργαλεία είναι πάρα πολύ σημαντικά ε, για την πλευρά της ενίσχυσης του μικρο, της μικροχρηματοδότησης. <clears throat> Äh, das Thema... Ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την μικροχρηματοδότηση, μικροδάνεια, το έχουμε συζητήσει πολύ στη Γερμανία και τα τελευταία 12 χρόνια στη μεταρρύθμιση κοινωνικής πολιτικής είχαμε τη δυνατότητα σε πολλούς ανεργούς να δημιουργήσουν μία εταιρεία ε, μοναδικού προσώπου, δηλαδή να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι και να ξεκινήσουν μία επιχείρηση με έναν απασχολούμενο. Ε, ήταν ένα πρόγραμμα αυτό και το οποίο ήταν πολύ πετυχημένο, ε, το οποίο λειτουργήσε μέσω των τοπικών οργανισμών εργατικού δυναμικού, ας πούμε των γερμανικών οργανισμών εργατικού δυναμικού και ε, αφορούσε κυρίως τεχνίτες οι οποίοι ε, μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς. Σε ορισμένους πέτυχε, μπόρεσαν να σταθεροποιήσουν, να σταθεροποιήσουν τη συμβολή τους στην αγορά, σε άλλους δεν πέτυχε. Όσον αφορά τώρα ε, το μέσον αυτό μπορέσαμε να διαθέτουμε 10.000 ευρώ σε σε, σε αυτά τα άτομα τα οποία ήταν αυτοαποσχολούμενοι αλλά επιχειρηματίες με την έννοια του μοναδικού προσώπου της εταιρεία ε, και 10.000 ευρώ και μπορέσαμε να τους βοηθήσουμε εν συνεχή να αναπτύξουν τις ε, δραστηριότητες τους. Ακούσαμε τώρα ότι υπήρχε η άποψη ότι αυτό αυτό το μέσον ήταν υπερβολικά περιορισμένο, υπερβολικά μικρό και αφορούσε, κάλυπτε πάρα πολύ μικρά προγράμματα και θα προτιμούσαν τότε τουλάχιστον να καλύψουν μεγαλύτερα προγράμματα, μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αλλά πιστεύω, δεδομένες ανεργίες θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε δυνατότητες ε, στους ε, τεχνίτες, στους αυτοαπασχολούμενους να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους και την αυτοαπασχόλησή τους με μικροδάνεια. Βεβαίω, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν υπάλληλοι κάπου, εργαζόντουσαν παλιότερα σε επιχειρήσεις και δεν ξέρανε, δεν είχαν ιδέα πώς να λειτουργήσουν μια δική τους επιχείρηση. Καταλαβαίνετε όταν κάποιος λοιπόν θέλει να αρχίσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα μόνος του πρέπει να έχει και τις απαραίτητες γνώσεις. Έπρεπε λοιπόν να εκπαιδευθούν, ε, να ενημερωθούν και για να μπορέσει να επιτύχει όλο αυτό το πρόγραμμα μικροχρηματοδότησης έπρεπε να φροντίσουμε και για την κατάλληλη κατάρτιση. Δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να οργανώσει και να κινηθεί μέσα στα πλαίσια μιας επιχείρησης. Διότι αν μόνο, δίναμε μόνο χρήματα θα το καταδικάζαμε σε αποτυχία. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσει αυτή η δυνατότητα, ιδιαίτερα σε περιφέρειες όπου το ποσοστό ανεργίας είναι πολύ ψηλό και στο μέλλον πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα έχει αποτελέσματα ε, αν δημιουργήσουμε και την κατάλληλη υποδομή ενημέρωσης και κατάρτισης για τους αυτοαποσχολούμενους και δι για τεχνίτες. Τώρα για τον τραπεζικό τομέα Στη Γερμανία έχουμε περιφερειακές ε, τράπεζες, ε, τράπεζες ε, που δίνουν στεγαστικά δάνεια, υποθήκες και λοιπά, τοπικές τράπεζες σε περιφέρειες, στα κρατήδια λοιπόν και αυτές οι μικρότερες τράπεζες οι οποίες κινούνται κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο ε, δεν ε, ε, υπέφεραν τόσο πολύ όσο οι μεγάλες ομοσπονδιακές τράπεζες και διεθνείς τράπεζες. Είχαν λοιπόν λιγότερες δυσκολίες και όταν εξετάζαμε την πράσινη βίβλο για τη συγχρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε πει ότι αυτός ο τομέας των περιφερειακών τραπεζών και μικρότερων τραπεζών θα πρέπει να αναγνωριστεί τότε δεν είχε αναφερθεί από την Κομισιόν, αλλά αναγνωρίσαμε ότι για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων, οι περιφερειακές αυτές τράπεζες παίζουν έναν τεράστιο ρόλο. Λοιπόν, μέσα στο, στα διαφορετικά ταμεία θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια πρόβλεψη για κατάρτιση και μαζί με τα, την μικροχρηματοδότηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η στήριξη και η επιβίωση των μικροτέρων περιφερειακών τραπεζών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους ομιλητές στον κατάλογο. Άρα δίνουμε ξανά το λόγο στους τρεις ομιλητές. Θα μπορούσα να προσθέσω κι εγώ μια γενική ερώτηση. Προσπαθούσα να καταλάβω εάν κάνουμε ένα κατάλογο των πιο σημαντικών προβλημάτων που αποτελούν εμπόδια στην ανάπτυξη των διευκολύνσεων μικροπιστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το πλαίσιο των αυξανόμενων αναγκών χρηματοδότησης ε, των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ποια θα ήταν τα πιο σημαντικά θέματα σε αυτό τον κατάλογο, Τι πιο σημαντικές δυσκολίες, τα πιο μεγάλα εμπόδια στην περαιτέρω επέκταση αυτού του θεσμού. Δεύτερη ερώτηση. Η μικροπίστωση σήμερα θεωρείται ως ευκαιρία να ενταχθούν περισσότεροι στον, στην αγορά απασχόλησης. Δεν αναφερθήκατε στις γυναίκες, αναφερθήκατε στους Ρωμά για παράδειγμα, αλλά ε, εδώ θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο επίλυσης των διαρθρωτικών προβλημάτων. Ο, ο θεσμός των μικροπιστώσεων. Δεν υπάρχουν άλλοι στον κατάλογο. Α, ποιος θέλει να απαντήσει. Α, έχουμε μια ακόμα ερώτηση. Ναι, μια ερώτηση και μια παρατήρηση. Αυτά. Δεν μιλάμε για τεράστια ποσά και θα πρέπει να κινούνται σε ένα θετικό περιβάλλον. Εάν οι δαπάνες και η όλη λειτουργία της χρηματοδότησης μετατραπεί σε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό άχθος, τότε δεν θα, δεν θα, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και δεν θα είναι προσφυλής, δημοφιλής ε, στους ενδιαφερόμενους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ορθολογικοποιήσουμε τη λειτουργία του, να είναι απαλλαγμένο από βαριά γραφειοκρατία και να το κάνουμε ε, ελκυστικό έτσι ώστε να γίνει αποδεκτή η προσφορά του τομέα από τους ενδιαφερόμενους και να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις. Θέλει κάποιος να απαντήσει, λέει πρόεδρο. Κύριο Έριξον, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μια ερώτηση αφορούσε τα ποσοστά αθέτησης του τομέα ή πόσες από αυτές τις απόπειρες επιβιώνουν, αν θέλετε. Η εμπειρία μας δείχνει ότι με βάση τους εταίρους μας 12-25% των παρόχων πιστώσεων τελικά χάνονται. Μάλλον πραγματοποιούν ζημίες. Αυτό είναι το ποσοστό σφάλματος, λέει ο μιλητής. Να το συγκεκριμενοποιήσω, λέει η κυρία Κράι. Ρώτησα για το ποσοστό αποτυχίας. Εάν γίνονται περισσότερα σφάλματα ή λιγότερο από ό,τι σε μεγάλα προγράμματα. Υποθέτω γίνονται λιγότερα από ό,τι τα μεγάλα προγράμματα στη διαφορετική πολιτική. Εγώ δεν ρώτησα ποιε επιχειρήσει επιβιώνω, αλλά ποιο είναι το ποσοστό σφάλματος. Επιτυχίες και αποτυχίες υπάρχουν, αλλά Α, περισσότερο με ενδιαφέρουν η λανσασμένη υπεξεργασία αιτήσεων και πόσα, σε τι ποσοστό απορρίπτονται, είναι εσφαλμένες οι αποφάσεις. I think Ειλικρινά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο λείπουν κάποια αριθμοί. Αν κατάλαβα σωστά, εννοείται όταν κάποιος ξεκινεί μια επιχείρηση ή επεκτείνει μια επιχείρηση με την στήριξη της μικροπίστωσης, εάν συνεχίζει να εφίσταται μετά από ένα χρόνο, αυτό εννοείται. Ε, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες στη διάθεσή μας. Υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί μικροπιστώσεων που συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες, αλλά όχι όλες. Έχουν τους πελάτες τους, οι οποίοι ξεκινούν μια επιχείρηση, την επεκτείνουν. Αλλά δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα συνεχίσουν να έχουν επαφές μαζί τους μετά από ένα χρόνο. Δεν ξέρω, Μαρία, αν μπορείς να το επιβεβαιώσει αυτό. Αυτό απαντά τελικά. Μάλλον αυτή ήταν η ερώτησή σας, κυρία Κρέλ. Όχι. Δεν... Ε, ίσως να μην πάρετε απάντηση, διότι εμείς ε, σκεφτόμαστε το, το ε, προσωρινό ποσοστό σφάλματος ε, με τα δημόσια κονδύλια που χρησιμοποιούνται και μετά γίνεται κατάχρηση και υπάρχει, υπάρχουν λάθη στις δημόσιε συμβάσει. Ίσως αυτό να μην σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μικροπιστώσει για να στηρίξουν τους οργανισμούς ε, μικροπιστώσεων. Ο κύριο Έριξον, το ποσοστό σφάλματος θα πρέπει να είναι μηδέν τότε. Διότι το μόνο που τη χάνει στήριξη, είναι μικροπίστωση για επιχειρήσει, ε, σύμφωνα με τον ορισμό για ποσά κάτω από 25.000. Άρα όλα ελέγχονται, το κάθε δάνειο ξεχωριστά, όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας ε, τη χάνουν ελέγχου. Καλά αυτά τα νέα, πολύ καλή απάντηση. Μπορείτε να συνεχίσετε. Τώρα οι άλλες ερωτήσει. ήταν για τη ζήτηση. Όταν βλέπουμε τα μέσα χρηματοδότησης, έχουμε κάποιους περιορισμούς γεωγραφικούς. Δεν μπορούμε να κατανέμουμε όλους τους πόρους σε μια χώρα, αλλά δεν υπάρχει και ισότιμη κατανομή ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχει μεγαλύτερη ίσως ζήτηση σε κάποιες χώρες όπως είναι η Ρουμανία για μικροπιστώσεις από ότι εμείς μπορούμε να παρέχουμε έχουν ήδη φτάσει στο όριο. Άλλε χώρε όπως η Ιταλία, Πολωνία, Γαλλία, Ισπανία, εκεί υπάρχει ψηλότερη ζήτηση από ό,τι θα μπορούσαμε εμείς να παρέχουμε με βάση τα όρια που έχουμε. Από την άλλη πλευρά, κάποιε χώρες δεν έχουν καθόλου ζήτηση από ό,τι βλέπουμε, γιατί βλέπουμε τη ζήτηση μέσα από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Ε, αλλά και σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν ε, ε τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης. Μια άλλη ερώτηση ήταν ε, σε σχέση με τους τύπους ενδιαμέσων που χρησιμοποιούνται για να φτάσουμε στους μικροδανειστές. Είπα ότι ο πρώτος ε, στόχος δεν είναι οι τράπεζες, ε, αλλά θέλουμε να έχουμε συνεργασία, ιδιαίτερα με τις συνεργατικές τράπεζες γιατί σε σύγκριση με άλλες τράπεζες αυτές οι συνεργατικές έχουν ε, πρόσβαση σε σε απόμακρες περιοχές, σε ε, αγροτικές ε, περιοχές όπου δεν λειτουργούν οι εμπορικές τράπεζες πια. Τώρα, στα εμπόδια, ένα σημαντικό στοιχείο που βλέπω εγώ είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο τύπου αγορά, αλλά πρέπει να υπάρχουν και ιδιώτες επενδυτές. Υπάρχουν εθνικά σχέδια για μικροπίστωσης ε, και αυτό δεν βοηθά μακροχρόνια στην ανάπτυξη αηφόρων ιδρυμάτων μικροχρηματοδότησης. Ε, Βραχυπρόθεσμα μπορεί να είναι σωστό, αλλά δεν δημιουργεί αγορές. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα σε πολλές χώρες. Άλλο πρόβλημα στην αγορά. Όταν τα επιτόκια είναι ψηλά στις μικροπιστώσεις, ε, αυτό μπορεί να είναι δυνάμει ένας κίνδυνος. Δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ε, υπάρχει κέρδος στον τομέα των μικροπιστώσεων. Παρόλο που βλέπουμε ότι η τιμή των πιστώσεων είναι ψηλή και υπάρχουν και ε, ανώτατα όρια σε κάποιες χώρες στα επιτόκια. Αλλά με μικροπιστώσεις, παροχή μικροπιστώσεων υπό την ε, μορφή μη τραπεζικής μικροπίστωσης υπάρχουν ψηλά λειτουργικά κόστη που πρέπει να καλυφθούν και στην τελική ανάλυση θα ε, είναι πολύ ψηλή τιμή της μικροπίστωσης. Η κυρία Ντεσρίβερ. Yes, will... Ευχαριστώ για το νέο κανονισμό. Πράγματι, όπως είπα και στην παρουσία μου, η πλατφόρμα τεχνικής βοήθειας, τεχνικής αρρωγής βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας Στόχος είναι να βοηθήσουμε τις αρχές να διαχειριστούν καλύτερα, να τους δώσουμε κίνητρα, να στηρίξουν τις μικροπιστώσεις και να φέρουν στην επιφάνεια το συγκεκριμένο θέμα στη συζήτηση με τις διαχειριστικές αρχές. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο λαμβάνουμε υπόψη μας πολύ συγκεκριμένα στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας. Um, Maybe as question and maybe uh, Ms. can Επίσης ε, για το αν είναι ευκαιρία η μικροπίστωση να έρθουν οι νέοι στις αγορές και μπορεί να συμπληρώσει και η κυρία Νόβακ. Έχουμε παραδείγματα και νέων που μπορεί να ωφεληθούν από τις μικροπιστώσεις αλλιώς δεν θα ήταν ικανοί να έχουν κάποιες ευκαιρίες, δεν είχαν την δυνατότητα να πάνε στα πιστωτικά ιδρύματα. Έχουμε το παράδειγμα της MicroStart εδώ στις Βρυξέλλες και κάποιων πολιτών νέων σαν παράδειγμα μια υποψηφία η οποία έπρεπε να έχει πάντα το παιδάκι της μαζί της, το μωρό της μαζί της και παρόλα αυτά μπόρεσε με τη συγκεκριμένη βοήθεια να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ξεκινήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα και άλλα παραδείγματα. Η κυρία Νόβακ. για, τις, ε, για τη βοήθεια προς τις επιχειρήσεις. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και στον τομέα της κατάρτισης, ιδιαίτερα για αυτούς που είναι άνεργοι για μια κάποια περίοδο και έχουν χάσει κάποιες δυνατότητες και ικανότητες που είχαν παλιότερα. Παράλληλα λοιπόν με τις υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις κάποιες ενδιάμεση δίνουν στους πελάτες τους την δυνατότητα κατάρτισης, εκπαίδευσης, προετοιμασίας και σε επίπεδο διοικητικής βοήθειας, διαχειριστικής βοήθειας και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό σε άλλες περιοχές του κόσμου όπως την Ασία ε, τα πράγματα είναι κάπως πιο απλά. Κάποιες παραδοσιακές δραστηριότητες διεξάγονται χωρίς θέματα διοικητικά, γραφειοκρατικά, θέματα ασφαλείας. Ενώ στις δικές μας χώρες όλα είναι διακανονισμένα και περίπλοκα. Και ένα ways of uh, creating um, uh, uh, Βασικός στόχος λοιπόν όταν κάποιος θέλει να αρχίσει μια επιχείρηση είναι πρώτα να έχει λύσεις και να οδηγηθεί στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης όπου είναι εφικτό και να μειωθεί ο λεγόμενος ανεπίσημος τομέας. Σχετικά με τις δυνατότητες τώρα μικροπιστώσεων για κάποιες ομάδες κοινωνικές ευάλωτες. Φυσικά και αυτό εδώ έχει μεγάλη σημασία. Αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβαση στα παραδοσιακά πιστοτικά ιδρύματα. Στη Γαλλία, σαν παράδειγμα, έχουμε 30.000 πελάτες σε δραστηριότητα Σε κάποιες φάσεις το 200 θέσεις απασχόλησης την εβδομάδα. Το 5% από τους πελάτες αυτούς είναι Ρωμά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τους αριθμούς, αλλά επίσης ένας μεγάλος αριθμός των νέων εποφελήθηκε από ένα πρόγραμμα για τις φτωχές περιφέρειες, μετανάστες ή παιδιά μεταναστών καλύτερα, και τους παρέχουμε ένα πακέτο το οποίο αφορά και την κατάρτιση σε κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεύτερον, τους παρέχουμε ακριβώς τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία μικροεπιχειρήσεων και τρίτον, το λεγόμενο coaching, το οποίο θα τους βοηθήσει να πετύχουν την προσπάθεια που αναλαμβάνουν. Τώρα για τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Είναι σαφές ότι οι μακροπιστώσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να αποσβέσουν το κόστος τους. Στις υποανάπτυξη χώρες κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει εύκολα. Γιατί μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους υψηλά επιτόκια Πολλές φορές ε, αυτό ε, αντιπροσωπεύει το 20 με 30% του συνολικού κόστους. Ενώ στην Ευρώπη κάτι τέτοιο για τους γνωστούς λόγους δεν είναι δυνατόν. Θυμάστε την παλαιά διάκριση ανάμεσα στην προτεσταντική λογική και την καθολική λογική. Στις προτεσταντικές χώρες ο κόσμος εξακολουθεί να πιστεύει ότι το υψηλό επιτόκιο είναι απαράδεκτο, δεοντολογικά. Γιατί είναι εφικτό στις υπόλοιπες χώρες. Γιατί τα επίπεδα χρηματοδότησης είναι πάρα πολύ χαμηλά και το κόστος του επιτοκίου είναι και αυτό χαμηλό ανεξαρτήτως του ύψους του επιτοκίου. Μικρά δάνεια, γρήγορη απόσβεση, αποπλήρωση μάλλον, Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας προβληματίσει στην Ευρώπη. Παίρνω το παράδειγμα της Γαλλίας πάλι. Όταν ζητάμε από τους πελάτες μας τα πληρώσετε 20%. Λένε ναι, έχει σημασία να έχουμε πρόσβαση στην πίστοση, παρά να έχουμε χαμηλά επιτόκια. Έχουμε διάφορες τράπεζες οι οποίες αναχρηματοδοτούν τη δραστηριότητά μας και μας λένε όχι. Γιατί αυτό θα είναι πάρα πολύ κακό για την εικόνα της τράπεζάς μας. Και δεν το δέχονται. Είναι αλήθεια ότι η κοινή γνώμη σε ένα κράτος πρόνοιας δεν είναι διατεθειμένο για μικροπιστώσεις με επιτόκια 20-30%. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και οι περισσότεροι από τους ενδιαμέσους, οι οποίοι θα πρέπει να συνδυάζουν από τη μία την κάλυψη του κόστους τους, την αποδοτική τους λειτουργία δηλαδή, και από την άλλη να μπορούν πάντα να εξυπηρετούν τους κοινωνικούς τους στόχους, συνήθως αυτό που κάνουν είναι να εξυπηρετούν περισσότερο τους κοινωνικούς στόχους και δευτερευόντως προσπαθούν να καλύψουν το κόστος λειτουργίας τους. και συγκεντρώνουν την προσοχή τους πολλές φορές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολλές φορές σε προγράμματα που δεν είναι κάτω από 25.000 ευρώ αλλά κάτω από 150.000 ευρώ και έτσι δεν έχουν το πρόβλημα να καλύψουν το κόστος λειτουργίας τους. Έχουν όμως δυστυχώς εγκαταλείψει αυτή την πελατεία τους η οποία κανονικά θα έπρεπε να είναι η φυσική τους πελατεία, η φυσική πελατεία των μικροπιστώσεων. Τέλος. Για τις τελευταίες σας ερωτήσεις ποια είναι τα βασικά θέματα που δημιουργούνται για την ανάπτυξη των μικροπιστώσεων. Σας μίλησα για τις τέσσερις ε, τάσεις. Είναι μια στρατηγική σφαιρική αυτές οι τέσσερις προτάσεις. Δεν μπορεί κανένας να προωθήσει ένα κομμάτι και να εγκαταλείψει τα άλλα γιατί αυτόματα θα δημιουργείται ένα εμπόδιο, θα ορθώνεται ένα εμπόδιο. Αυτό το οποίο έχει σημασία για μένα είναι πρώτον να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει και η κοινή γνώμη, η άποψη της κοινή γνώμης. Έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά θεωρεί, εξακολουθεί να θεωρεί, ότι η Ευρώπη είναι μια περιφέρεια όπου ο κόσμος περισσότερο θα πρέπει να λειτουργεί με έμιστη εργασία και αυτοί οι οποίοι δεν απασχολούνται με τον τρόπο αυτό θα πρέπει απλά να τύχουν βοήθειας. Έτσι λοιπόν, για να ανάξει ο νόμος πρώτα απαιτείται να, να αλλάξει η αντίληψη. Και για να αλλάξει η αντίληψη του κόσμου σημαίνει ότι απαιτείται πολλή επικοινωνία, πολλή ενημέρωση, χρηστές πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και στο ίντερνετ και με πολλούς άλλους τρόπους. Αυτό έχει σημασία. Εμείς δεν βρισκόμαστε σε μία παρούσα φάση κρίσης απλά, αλλά σε μία παρούσα φάση η οποία χαρακτηρίζεται από τη βαθιά αλλαγή της οικονομίας. Και γι' αυτό δεν θα πρέπει να χάσουμε το πλεονέκτημα που είχαμε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αλλαγές. Οι Πρόεδρος, δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, οι ομιλητές θέλουν να λάβουν το λόγο, οι άλλοι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, διότι πιστεύουμε ότι αυτή την πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε να προχωρήσει η Ευρώπη προς μια ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη και επίσης να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλλει και η πολιτική συνοχή από τη βάση στην οικονομική μας ε, ανάπτυξη και ευημερία. Ε, πιστεύουμε ότι όλο αυτό το πλαίσιο της πολιτικής συνοχής μπορεί να προσφέρει περισσότερα ε, και μπορεί να αναπτυχθεί έτσι ώστε να στηρίξει και τον τομέα της μικροχρηματοδότησης είσαστε πιστεύω μόνος φορέας ε, με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, να διαβουλευτούμε και η Κομισιόν σίγουρα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της. Όμως τα μεμονωμένα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία ακόμα προσφέρουν το νομικό πλαίσιο της, ε, ε, στον τομέα αυτών και ιδιαίτερα στις μικρότερες χώρες ε, αυτός ο τομέας της μικροχρηματοδότησης ε, θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο μέλλον ε, και όταν συζητιούνται στην Κομισιόν τα εταιρικά προγράμματα και τα εταιρικά προγράμματα συνεργασίας συνεργασίες λαμβάνουν λαμβάνονται υπόψη ακριβώς και αυτός ο τομέας της μικροχρηματοδότησης. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσουμε τώρα αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξή μας και είμαστε και στην ώρα μας για να προχωρήσουμε στο σημείο 5. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε με το σημείο 5 η Κομισιόν είναι εδώ. Έχουμε τη, τον κατεξουσιοδότηση κανονισμό να συζητήσουμε. Να σας ενημερώσω σύντομα ότι αυτός ο κανονισμός πέμφθηκε στο Κοινοβούλιο στις 3 Μαρτίου και διαναμήθηκε αμέσως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τη Γραμματεία και η προθεσμία των δύο μηνών που είχαμε να προβάλλουμε αντιρρήσεις είναι από τις 7 Μαρτίου και για το Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 7 Μαρτίου με 7 Μαΐου. Μπορούμε να ζητήσουμε βεβαίως και την παράταση αυτή των δύο μηνών. Και σας θυμίζω, αν εμείς ως Επιτροπή Ρέτζι ε, φέρουμε αντίρρηση σε αυτές τις ε, πράξη κατά εξουσιοδότηση, τότε χρειαζόμαστε ένα ψήφισμα το οποίο θα πρέπει να παρουσιαστεί και να ψηφιστεί στην επόμενή μας συνεδρίαση στην 1η Απριλίου και συνεχεία να ε, περιληφθεί στην ατζέντα της, μάλλον της δεύτερης Ολομέλειας του Απριλίου. Αυτός λοιπόν είναι ο, η διαδικασία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε στείλει το σχέδιο ε, το σχέδιο έξεση σε όλους δεν έχουμε λάβει αντιρρήσεις προς το παρόν προς τον, τον κανονισμό τα κατεξουσιοδότηση θα κάνουμε λοιπόν τη συζήτηση σήμερα και υπάρχει ευκαιρία να δούμε αν υπάρχουν αντιρρήσεις να καταγράψουμε τις αντιρρήσεις αυτές και εν συνεχεία να προχωρήσουμε στη σύνταξη ενός σχεδίου ψηφίσματος και όπω σα είπα μετά το ψήφισμα πρέπει να πάει στην Ολομέλεια. Ε, στο τέλος της συζήτηση θα καταλήξουμε στην ε, προθεσμία, καταληκτική προθεσμία υποβολής και εάν δεν γίνουν όλα αυτά τότε ο ρόλος της Επιτροπής μας ε, σταματάει σε αυτό το σημείο και ο κανονισμός πλέον ε, εφαρμόζεται, υλοποιείται μετά από τους δύο μήνες προθεσμίας. Η Κωνσταντσα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία τα είπατε. Ε, επί της διαδικασίας εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι ήδη το Δεκέμβριο συζητήσαμε την πρώτη έκθεση του κατεξουσιοδότηση κανονισμού ε, και ε, είχαμε, οργανώσαμε στο μεσοδιάστημα ορισμένες ε, συναντήσεις να συζητήσουμε αυτόν τον κανονισμό. Αυτός ο κανονισμός τώρα συντίθεται από διάφορα τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν όλα συγκεραστεί κάτω από έναν κατοξουσιοδότηση κανονισμό ο οποίος όμως δεν είναι και κατεπήγον, να μετατραπεί δηλαδή σε νομικό μέσο για να υλοποιηθούν τα λειτουργικά προγράμματα και να υλοποιηθούν οι στόχοι της συνοχής. Δηλαδή τι εννοώ, ότι ίσως δεν έχετε όλοι μελετήσει αυτόν τον ε, κανονισμό κατεξουσιοδότηση Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω ορισμένα παραδείγματα Παραδείγματο χάρη ε, χρηματοδοτικές διορθώσεις, ορισμένες διατάξεις ε, για τα χρηματοδοτικά μέσα, μέσα στο πλαίσιο των ε, χρηματοδοτικών ε, οργανισμών, παραδείγματο χάρη κάλυψη κόστους ε, ταξιδίων, στέγασης, κάλυψη του στόχου των δοκιμών. Ε, είναι δηλαδή ακριβώς ε, καλύπτει τεχνικά όλα τα ζητήματα τα οποία έχουμε εμείς αποφασίσει στο βασικό κανονισμό. Καλύπτει όλες τις τεχνικές πτυχές εμείς είχαμε συζητήσει και εις βάθος ορισμένα επιμέρους ζητήματα. Και το πιο καυτό ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αυτά τα τρία παραρτήματα. Αυτά τα τρία παραρτήματα τα οποία ε, είχαν συναυθεί στον ε, κατεξουσιοδότηση κανονισμό. Μάλιστα στο τελευταίο παράρτημα υπάρχουν ένα σωρό στοιχεία ε, στην, στο πρώτο σχέδιο του κανονισμού ε, είχαμε αναγκαστεί να αντιμετωπίσουμε πάνω από 100 σελίδες ερωτημάτων από τους ενδιαφερόμενους ε, και σήμερα θα θέλαμε να, να ξέρουμε εάν η Κομισιόν μπορεί να μας εξηγήσει γιατί δεν κατάφεραν αυτών των αριθμών των ερωτήσεων των εκκρεμών ζητημάτων να τα μειώσουν περαιτέρω Δυστυχώς, μόνο την περασμένη εβδομάδα τέθηκε το ερώτημα εάν θα πρέπει οι αλληλείς των ωκεανών ή των ε, βαθυπαλλαγικών ψαριών και οι, αλλοί, και οι, ψα, ε, ερασιτέχνες ψαράδες που ψαρεύουν στις εσωτερικές λίμνες και λιμνούλες να καλυφθούν από το ίδιο παράρτημα και γιατί δεν μπόρεσαν να μειώσουν λοιπόν όλες αυτές τις λεπτομερείς ε, πτυχές. Συζητήσαμε με μακρόν με τους εισηγητές αλλά και με τους σκιώδεις εισηγητές και δεν είδα να υπάρχουν αντιρρήσεις ε, για τον κανονισμό αυτό και δεν υπάρχει μια ισχυρή βούληση απόρριψης του κανονισμού. Συνάγω λοιπόν ο Τσιμπερένο ότι υπάρχει μια ευρεία συνένεση για τον κανονισμό αυτό. Απλώς ε, θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν ε, τι θα γίνει εάν τυχόν προτείνουμε μια διαφορετική νομική βάση. Πιστεύω ότι το νωρίτερο που μπορεί να υποβληθεί θα είναι το Σεπτέμβριο δηλαδή στη νέα θητεία του νέου σώματος, οπότε πάμε προς το τέλος του τρέχοντος έτους, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Δεδομένου ότι ακόμα θα καταβληθούν πιστώσεις φέτος. Και άλλα, όχι μόνο αυτό, θέλουμε να ξεκινήσουμε το ταχύτερο στην υλοποίηση προγραμμάτων ε, στο να ξεκινήσουν η εκτέλεση συγκεκριμένων έργων και αν δεν υπάρχει η νομική βάση για τα εκτελεστικά προγράμματα θα παρουσιαστεί ένα τεράστιο φρένο στην εξέλιξη και στην υλοποίηση των προγραμμάτων, το οποίο θα ήταν απαράδεκτο για τις περιφέρειες πιστεύω ότι ήδη στην υπερψήφιση του γενικού κανονισμού, του βασικού κανονισμού, είχαμε δείξει ότι έχει διαγραφεί ένα μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος και υπάρχει μια γενική αποδοχή ότι όλα τα ταμεία αυτά θα πρέπει να εμπίπτουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο, το οποίο είναι προς όφελος της ε, μείωσης της γραφειοκρατίας. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τα σχόλια της Κομισιόν για τα παραρτήματα, αλλά σας παρακαλώ θερμά εδώ να εγκρίνουμε ως Κοινοβούλιο τον, ε, τους ε, κατεξουσιοδότηση κανονισμούς αυτούς και χωρίς αλλαγή και να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να δράσει γρήγορα, δεδομένου ότι βρισκόμαστε, βρισκόμαστε υποχρονική πίεση και πρέπει από κοινού να καταλήξουμε σε μία απόφαση σε αυτόν τον, τον τομέα. Ευχαριστώ. Να δώσω τον λόγο στο Λάμπερτ εν συντομία και ε, Νίκολα θα πρέπει να μας πείσει τελικά για τα στοιχεία. Ευχαριστώ να προσθέσω κάτι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ε, υλοποίηση όλων αυτών των συζητήσεων και αρχών που έχουμε αποδεχτεί στο γενικό κανονισμό και έχουμε και από την άλλη πλευρά τον ε, κατεξουσιαδότηση κανονισμών που είναι πολύ λεπτομερής. Ερώτηση προς την Κομισιόν από μέρους μου. Μπορούν να μας πούν ποια θα μπορούσε να ήταν η επίδραση ή το αποτέλεσμα εάν είχαμε μια νέα συζήτηση για τις λεπτομέρειες. Υπάρχουν πολλοί άριθμες σελίδες εδώ μπροστά μας. Ποια είναι η επίδραση της έναρξης των νέων προγραμμάτων. Πρώτη ερώτηση αυτή. δεύτερη. Μπορεί να μας δώσει η Κομισιόν κάποια στοιχεία σχετικά με την συζήτηση που έχει πραγματοποιηθεί στο Συμβούλιο Έχω κάποιες πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι το Συμβούλιο έχει επίσης ζητήσει μείωση όλων αυτών των λεπτομερών ερωτήσεων. Και τρίτον, θα μπορούσε να μας πει η Κομισιόν ποιος πρέπει να εκπληρώσει όλα αυτά τα στοιχεία και τα νούμερα. Έχω την εντύπωση ότι οι αποδέκτες, οι, για παράδειγμα οι αγρότες ή οι αλλοίς, πιστεύουν ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν οι ίδιοι όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτό μπορεί να γίνει αυτόματα σε επίπεδο έργου ή είναι μια παρανόησή μου. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ε, η Ιβέρς δεν είναι εδώ. Η Ελίζαμπετ θα ήθελε να μιλήσει. Ναι. Και εγώ επανέρχομαι στα παρατήματα όμως εμένα με ενδιαφέρει η συνοχή των παρατημάτων αυτών με την εφαρμοστική πράξη η οποία παραπέμπει στα στοιχεία. Τώρα, έχουν συντμηθεί τα παραρτήματα έναντι της αρχικής έκδοσης και Υπάρχει αυτή η συνέπεια, αυτή η συνοχή με τα προηγούμενα ή υπάρχουν στοιχεία ε, στα παρατήματα στα οποία δεν μπορούμε καθόλου να εκφράσουμε την άποψή μας. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Δηλαδή, θα μπορούσα να δεχτώ αυτόν το, αυτούς τους κανονισμού εφόσον συνάδουν με την εφαρμοστική πράξη, με τον εφαρμοστικό κανονισμό ε, και εφόσον δεν περιορίζουν την δική μας ε, δυνατότητα παρέμβασης. Αλλά εάν τώρα αυτό το παράρτημα διαφέρει μεταξύ της εφαρμοστικής πράξης, ε, τότε όσοι προετοιμάζουν τα προγράμματα θα βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Αυτό είναι το βασικό μου ερώτημα. Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία ακούστηκαν από τους συναδέρφους, γιατί πολλά από τα σχόλια αυτά θα μπορούσα να τα κάνω κι εγώ. Απλά θα ήθελα κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τις δημοσιονομικές διορθώσεις και πώς μπορούμε να κάνουμε τις διορθώσεις αυτές και τις ε, ε, μεταβατικές περιόδους που είναι απαραίτητες για τα ελεγκτικά όργανα έτσι ώστε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργούν σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες. Πρέπει να υιοθετηθεί αυτή η πράξη, αλλά θα πρέπει να ε, ξεκαθαριστούν οι κανόνες. Κορνέλια, έχεις το λόγο για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Ο Γιώνας είναι σκιώδης εισηγητής και επειδή το θέμα είναι περίπλοκο έχω ένα ερώτημα στο άρθρο 3. Όσον αφορά αυτές τις ε, δημοσιονομικές διορθώσεις, το ΑΒΓ τα καταλαβαίνω, αλλά τι σημαίνει τώρα λεπτομερός. Ε, τι σημαίνουν, τι νόημα έχουν αυτές οι διατάξεις λεπτομερώς, ε, υπάρχει κάποια δυνατότητα κλιμάκωσης, υπάρχουν άλλα στοιχεία ε, τα οποία λείπουν, θα ήθελα κάποιες επεξηγήσεις επί του άρθρου 3. Όπως σας είπα, η συζήτηση που έγινε μεταξύ των σκιωδών εισηγητών δεν την παρακολούθησα. Ευχαριστώ βέβαια. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα ήθελα να θίξω ένα ουσιαστικό σημείο. Πιστεύω ότι με την περιφερειακή πολιτική τώρα έχουμε καταλήξει σε μια ολοκλήρωση σημαντική της, ε, των νομικών εργασιών η οποία τράβηξε επί χρόνια και έτσι μπορούμε να πούμε και στις εκλογικές μας εκστρατείες ότι έχουμε ενισχύσει κατά πολύ ε, το, νομικό πλαίσιο στήριξης των περιφερειών. Όμως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και το θέμα που με απασχολεί εμένα είναι στο τιμίο αλίας. Όπως είπε και η συνάδελφός μας, ε, όσον αφορά την, την ε, ε, αλία στους ωκεανούς και την αλία σε, σε λίμνες, όλα αυτά τα έχουμε μαζέψει και πακετάρει υπό ένα παράρτημα. Δεδομένου ότι αυτή η εργασία απασχολεί και το ελεγκτικό συνέδριο και δεδομένου ότι θέλουμε να μειώσουμε την γραφειοκρατία, καταλαβαίνω ότι θέλουμε να συγκεράσουμε τους δύο ακραίους πόλους, ωκεανούς και λιμνούλες, αλλά ε, για την μικρή αλληλεία, για τις μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να ε, είμαστε βέβαιοι ότι οι προτάσεις ε, είναι σωστές και ότι εμπίπτουν σε ένα σωστό πλαίσιο για να δώσουμε και να μήνυμα στους πολίτες ότι κάθε φορά που παρουσιάζονται τέτοιες λεπτομέρειες σε τόσο πολλά έγγραφα και σελίδες δεν χάνουμε τον μπούσουλα όπως λένε και ότι ξέρουμε τι κάνουμε. Νίκολας, το μέλλον είναι στα χέρια σου θα πρέπει να μας πείσεις γιατί οι χρονικές προθεσμίες είναι μικρές. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία θέσατε. Εγώ θα βασιστώ στο παράρτημα 3 με όλα τα δεδομένα και τις χρηματοοικονομικές, δημοσιονομικές συγγνώμη διορθώσεις. Αυτό έχει σημασία. Καταρχάς, έχει προηγηθεί, όπως είπα, διαβούλευση, ιδιαίτερα για την κατεξουσιοδότηση πράξη σχετικά με τον κανονισμό των κοινών προβλέψεων και ρυθμίσεων. Ξεκινήσαμε εδώ και αρκετό καιρό, γιατί χρειαζόταν χρόνος. Οι πρώτες συζητήσεις έγιναν στα μέσα του προηγούμενου χρόνου. Έγιναν 15 επαφές με εμπειρογνώμονες από διάφορα κράτη-μέλη και οι τελευταίες συναντήσεις ήταν οι επίσημες για την προετοιμασία της κατεξουσιοδότησης πράξης, ε, ενεπλάκη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος αυτής της διαβούλευσης εκ των προτέρων ήταν να εντοπίσουμε τα προβληματικά θέματα. Όλοι θα θέλαμε να έχουμε στη διάθεσή μας μια κατεξουσιοδότηση πράξη, η οποία δεν θα δημιουργήσει αντιθέσεις, δεν θα επιβάλλει εμπόδια, και θα είναι απολύτως τεκμηριωμένη. <clears throat> Στα πλαίσια της συνάντησης των εμπειρογνωμόνων συγκεντρώσαμε την προσοχή μας στο παράρτημα 3, στο Άνεξ 3. Εκεί έγιναν τα περισσότερα σχόλια από τους εκπροσώπους των κρατών μελών. <clears throat> Αν πάμε λίγο πίσω και δει κάποιες περισσότερες προτάσεις ε, θα δει ότι το παράρτημα ήταν μεγαλύτερο από ό,τι είναι τώρα. Ξεκαθαρίσαμε λίγο τα πράγματα. Είχαμε 135 τομείς στο παράρτημα 3 και τώρα είμαστε στους 113. Προσπαθήσαμε λοιπόν και εγώ προσωπικά έκανα κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να αφαιρέσω ότι δεν είχε μία ξεκάθαρη τεκμηρίωση τεκμηρίωση σχετικά με τις ανάγκες που έχει η διαχειριστική αρχή για να φέρει σφαίρα στην αποστολή της. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια παρανόηση για το ποιος είναι αυτός που θα δίνει τα δεδομένα, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα συμπληρώνει τα δεδομένα. Αυτό το οποίο μιλάμε εδώ είναι το σύστημα ελέγχου ε, το ηλεκτρονικό, το, το πληροφορικό, το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί και να ελέγχεται από τη διαχειριστική αρχή. Εμείς εδώ ε, καθορίζουμε τον ελάχιστο ε, αριθμό πεδίων το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείτε. Όταν η διαχειριστική αρχή λοιπόν καθορίσει το σύστημα αυτό το πληροφορικό, τότε θα πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχει η δυνατότητα input για όλους αυτούς τους τομείς. Όχι για τους ε, άμεσους ωφελημένους, τους πολίτες, τους μεμονωμένους, τις μικρομεσαίες. Αυτοί είναι τομείς δεδομένων χρήσιμη για τη διαχειριστική αρχή και καλύπτει και τα τρία ταμεία. Γιατί τώρα πλέον έχουμε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου διαχειριστικό και για το κοινωνικό ταμείο και για το ταμείο συνοχής και το IMFF. E καλύπτει λοιπόν και τα τέσσερα εισαγωγικά ταμεία. Όπως είδατε κάποια από τους, κάποιοι από τους τομείς αυτούς αφορούν ένα μεμονωμένο ταμείο δεν είναι κάθε τομέας για όλα τα ταμεία, αυτό ξεκαθαρίζεται. Συμπληρωματικά ένα κράτος μέλος μπορεί να πάρει την απόφαση που καθιστά κάποιους άλλους τομείς ε, να μην έχουν σημασία. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό, αλλά λέμε, ας υποθέσουμε, ότι εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο επιδίωξης απλούστευμένου κόστους. Τότε δεν τίθεται το θέμα ύπαρξης του συγκεκριμένου πεδίου. Το πεδίο υπάρχει εκεί δηλαδή όταν είναι εφαρμόσιμο όταν μια χώρα κάνει επενδύσεις με τον τρόπο με τον οποίο απαιτεί τα δεδομένα αυτά να διορθωθούν. Τα δεδομένα αυτά πιστεύουμε ότι χρειάζονται για τη διαχειριστική αρχή να φέρει εις πέρα στις υποχρεώσεις της και να αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι και εμείς να αναφερθούμε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Για τα χρηματοδοτικά μέσα σαν παράδειγμα ενισχύσαμε τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε τις λεπτομέρειες και να συγκρίνουμε και να κάνουμε συμβατά τα δεδομένα που έχουμε στο CPR έτσι ώστε να παρακολουθούμε από κοντά το τι ακριβώς ε, συμβαίνει με τα χρηματοδοτικά μέσα. Ε, σχετικά με τους δείκτες επίσης, χρειάζεται ε, να είμαστε ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα προγράμματα, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δίνουμε πληροφορίες για τους προσανατολισμούς των τελικών αποτελεσμάτων προς τα τελικά αποτελέσματα με βάση τους δείκτες. Το πλαίσιο επίδοσης εξαρτάται από το αν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα και κατάλληλοι δείκτες. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται μεταξύ τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλα όσα βρίσκονται εδώ είναι τεκμηριωμένα, είναι συμβατά με το τι έχουμε στις εφαρμοστικές πράξεις και στη συγκεκριμένη αυτή ε, κατεξουσιοδότηση πράξη καθορίζουμε το ελάχιστο επίπεδο ε, ε, πληροφορικής ρύθμισης, ελέγχου και διασφαλίζουμε νομίζω την συμβατότητα ανάμεσα στους διάφορους τρόπους ελέγχου. Υπάρχει επίσης και το λεγόμενο e-cohesion ηλεκτρονική, ε, ε, ε, κάτι το οποίο θα ωφελήσει στους δίχεουχους να έχουν όχι την υποχρέωση αλλά την δυνατότητα να δίδουν στοιχεία στις αρμόδιες αρχές με ηλεκτρονικό τρόπο. Ηλεκτρονική συνοχή λοιπόν. Όταν ένας δικαιούχος κάνει μία έκθεση, παρουσιάζει ε, μια αίτηση χρηματοδότησης, μπορεί να το κάνει online, δεν πρέπει να το κάνει με ένα χαρτί και αυτό απλουστεύει τις διαδικασίες. Τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν ένα μέσο ηλεκτρονικό ε, στον τομέα της συνοχής, το οποίο να είναι συμβατό με το σύστημα πληροφορικής το οποίο είναι υποχρεωμένοι να διαχειρίζονται. Έτσι ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν online να έρχονται και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του συστήματος. Για το Ταμείο Αλίας τώρα. Στον τομέα της Αλίας, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Υπογραμμίζω ότι εδώ δεν ασχολούμεθα με τον Αλιέα, με τον πολίτη. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να μην είναι ειδικά για τον συγκεκριμένο πολίτη, Αλιέα, αλλά για την διαχειριστική αρχή. Όταν τα κράτη-μέλη δημιουργούν το σύστημά τους, θα πρέπει το σύστημα αυτό να είναι σε θέση να δώσει τα προαπαιτούμενα και να συλλέγει όλες τις πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται για όλα τα προγράμματα και για τα τέσσερα ταμεία. Για τις ε, διορθώσεις σχετικά με το πλαίσιο επίδοσης. Αυτό το οποίο εδώ ρυθμίζεται στον κανονισμό είναι ότι κλείνει ένα πρόγραμμα όταν δεν ε, επιτευχθούν οι στόχοι, υπάρχει απόκληση από τους στόχους, τότε θα πρέπει να υπάρξουν οικονομικές ε, ε, διορθώσεις. Καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι διορθώσεις αυτές και ο μηχανισμός ο οποίος δημιουργείται έχει σαν στόχο να συνδέεται το επίπεδο της υποεπίδοσης με το επίπεδο της διόρθωσης. Όχι κάθε φορά να αποφασίζουμε κατά περίπτωση δηλαδή το τι θα κάνουμε. Αυτό θα δημιουργήσει μια αβεβαιότητα. Θέλουμε λοιπόν κάποιους κανόνες οι οποίοι να συνδέουν τα προβλήματα που έχει ένα πρόγραμμα σε σχέση με την απορροφητικότητά του σαν παράδειγμα και ο δείκτης αυτός της υποαπορροφητικότητας συνδέεται με την δυνατότητα παρέμβασης και διόρθωσης. Για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας λοιπόν κάποιες δυνητικές δυσκολίες και ανομαλίες για τη λειτουργία ενός αυτόματου συστήματος πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όπου πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την αναλογικότητα το επίπεδο διόρθωσης μειούται και αυτό μας δίνει αυτή την ευελιξία που χρειαζόμαστε να έχουμε μία δυνατότητα διόρθωσης η οποία να είναι τεκμηριωμένη σε κάθε περίπτωση. Για τις άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν ε, σχέση με σημαντικές ελλείψεις οι οποίες ε, σημειούνται, η ελεγκτική διαδικασία η οποία εφαρμόζεται σήμερα καθορίζει το πότε υπάρχει μια βασική ε, απόκληση και πόσο σοβαρή είναι η απόκληση αυτή και έτσι καθορίζεται και αναλογικά το επίπεδο διόρθωσης. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είναι επίγον όλοι αυτοί οι κανόνες να τεθούν σε λειτουργία γιατί είναι κρίσιμοι για τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να δημιουργήσουν τα συστήματά τους και να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά τα συγκεκριμένα προγράμματα. Τα κράτη-μέλη όταν δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστημά τους στο IT, τότε προφανώς τα πράγματα δυσκολεύουν και σε σχέση με τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει το σύνολο των κανόνων να είναι διαθέσιμο άμεσα γιατί αυτό θα χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη για να προπαρασκευαστούν για την δημιουργία των χρηματοδοτικών μέσων των δικών τους, για τον καθορισμό των ελεγκτικών αρχών των δικών τους και αν όλα αυτά δεν είναι διαθέσιμα εκ των προτέρων δεν θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν με τον δικό τους προγραμματισμό. Εάν δεν ορίσουμε από τώρα την μεθοδολογία τότε και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπής και από πλευρά κρατών μελών θα υπάρξουν μπλοκαρίσματα. Αν υπάρξει δηλαδή αδυναμία έγκρισης της κατεξουσιοδότηση πράξη και εφαρμογής της κατεξουσιοδότηση πράξη άμεσα πριν από, από τον τερματισμό της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής εντολής τότε θα καθυστερήσουμε τα προγράμματα κατά έξι τουλάχιστον μήνες. Δεν απάντησε στην ερώτηση της Μπέδη για την συνέπεια ανάμεσα στις πράξεις. Ναι, είχα αναφερθεί να υπογραμμίσω ότι υπάρχει κάποια διάρθρωση ανάμεσα στο τι υπάρχει στο παράρτημα 3 της κατεξουσιοδότηση πράξης και κάποιων εκτελεστικών πράξεων, όπως κατηγορίες παρέμβασης, και ε, έχουμε ελέγξει την συνέπεια. Δεν υπάρχουν κάποιες ασυνέχειες και ασυνέπειες ανάμεσα σε αυτά, εξ όσων γνωρίζουμε. Και πρέπει, οπωσδήποτε, να υπάρχει συνέπεια. Είναι μία από τις προκλήσεις αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, Κάποιοι από αυτούς τους λεπτομερείς ε, κανονισμούς βρίσκονται σε εξουσιοδότηση πράξη, σε εκτελεστική πράξη, διαφορετικές διαδικασίες, διαφορετικό το timing. Αλλά οι μόνες εκτελεστικές που είναι οριστικοποιημένες είναι αυτές ε, σχετικά με την κατηγορία των παρεμβάσεων. Οι περισσότερες εκτελεστικές αυτή τη στιγμή περνάνε από τη διαδικασία της επιτροπολογίας πρέπει να οριστικοποιήσουμε τις κατεξουσιοδότηση πράξεις έτσι ώστε να τις ε, εναρμονίσουμε και να σε ευθυγραμμίσουμε με το υπόλοιπο κείμενο, έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια όντως. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια, Ελίζα Πέτ. Θέλω να θέσω το ερώτημα συγκεκριμένο Ε, από την πλευρά εκείνων που πρέπει να εφαρμόσουν, να υλοποιήσουν τα θέματα. Αυτά που μας είπατε σημαίνει ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν περικοπεί, συντμηθεί, έναντι του αρχικού σχεδίου, ότι αυτά που κόπηκαν δηλαδή, είναι όλα τα στοιχεία ή βάση του εφαρμοστικής πράξης υπάρχει και άλλη μια κατηγορία δεδομένων που εάν θα, θα επανέλθουν ε, στην, ε, στον κατοξουσιοδότηση κανονισμό παρόλο που κόπηκαν στα παραρτήματα. Υπάρχει δηλαδή θα ξεφυτρώσουν και άλλα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιληφθούν στο κανονισμό. Ευχαριστώ ο κύριος ε, Τσέλερ. Η Κομισιό μας είπε ότι ο κανονισμός αυτός τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον κανονισμό πλαίσιο, έχει μια ουσιαστική σημασία. Και έτσι λοιπόν ε, δεν καλύπτει μόνο τις δικές μας αρμοδιότητες, είναι άλλωστε και ε, συναρμόδια η Επιτροπή ε, Απασχόλησης, για τη γνωμοδότηση δηλαδή. Ε, και ιδιαίτερα ε, μα απασχολεί το θέμα της, ε, του, του, του Ταμείου Θαλάσσης και Αλίας. Ρωτώ λοιπόν, όπου υπάρχουν και τα προβλήματα, ρωτώ λοιπόν εάν έχουν συμφωνηθεί όλα τα δεδομένα σε αυτό το τομέα, σε αυτό το ταμείο. Δεν θέλω να συνενέσω σε κάτι και αργότερα να με δίρουν γι' αυτό. Χωρίς να είμαι βέβαιος ότι όσοι είναι αρμόδιοι και εμπειρογνώμονες αυτού του τομέα έχουν προηγουμένως συμφωνήσει και συνενέσει. Εάν δεν συμφωνήσουμε τώρα, θα καθυστερήσουμε έξι μήνες. Αυτό δεν με τρομάζει εμένα ιδιαίτερο με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Νομίζω ότι καλό θα μας κάνει να έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να επεξεργαστούν ή να προχωρήσουν περισσότερο στις εταιρικές τους συμφωνίες κλπ. Ε, και να μπορέσουν να συγκεράσουν τις εκτελεστικές τους δομές, ε, να μελετήσουν νέα προγράμματα κλπ και αν δω τώρα από την επιστολή της Προέδρου μας ε, ε, τα δεδομένα για το 2015, μελλοντικές πληρωμές κλπ, προτεραιότητα έχει η πληρωμή προηγουμένων προγραμμάτων του προηγουμένου έτους και όχι η πληρωμή, η καταβολή δηλαδή των αναγκαίων κονδυλίων για τα προγράμματα του επομένου έτους. Άρα λοιπόν δεν μας καίει, δεν μας πειράζει και τόσο πολύ μία καθυστέρηση. Απλώς θέλω να είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι ε, γνωρίζουν αυτό τον κανονισμό ενδελεχώς από τον ε, τομέα το, ε, αλίας και των θαλασσών για να μην μπλέξουμε στο μέλλον σε χειρότερα. Έχουμε ήδη απο... πάρει απάντηση από την Επιτροπή ότι δεν έχουν οποιαδήποτε αντίρρηση ε, σε αυτή την απάντηση. Άλλε ερωτήσει, όχι. Νίκολα μπορεί να κάνει τη δική σου τελική δήλωση. Ευχαριστώ. Να επανέλθω σε αυτό το σημείο σχετικά με τις εκτελεστικέ πράξεις. Υπάρχουν δύο ξεχωριστά πράγματα. Στην κατεξουσιώδηση πράξη έχουμε τι ελάχιστε προποθέσει σε ό,τι φορά τα συστήματα πληροφορικής που πρέπει να έχουν οι διαχειριστικέ αρχές και τι δεδομένα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν. Μέσω εκτελεστική πράξη δεν θα κάνουμε κάτι που να προσθέσει σε αυτά. Δεν μπορούμε. Δεν θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Και δεν θα συμβεί. Αυτό που καθορίζεται σε αυτό το παράρτημα είναι το κατάλογος των των απαιτούμενων δεδομένων. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να προσθέσει φυσικά περισσότερα παιδεία, αν το θέλει, αν θεωρεί ότι διευκολύνει τον τρόπο διαχείρισης ενός προγράμματος. Αλλά σε ό,τι φορά τα υποχρεωτικά παιδεία, του συστήματος πληροφορικής. Αυτά καθορίζονται στην κατεξουσιοδότηση πράξη. Δεν θα προσθέσει ε, οποιαδήποτε εκτελεστική πράξη οτιδήποτε άλλο. Τώρα, ε, στο θέμα του timing, για να απαντήσω στον κύριο Τζέλερ. Ε, δεν ε, θα συμφωνούσαμε ότι δεν έχει σημασία αν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Σίγουρα θα στείλει ένα αρνητικό μήνυμα εάν δεν καταφέρουμε να οριστικοποιήσουμε το νομοθετικό πακέτο τώρα. Και πιστεύουμε ότι ε, πρακτικά, εάν δεν υπάρχει το πλαίσιο, θα επηρεάσει αρνητικά τα κράτη-μέλη, καθώς αυτά προσπαθούν να ξεκινήσουν την υλοποίηση των προγραμμάτων. Ελπίζουμε φυσικά ότι τα πρώτα προγραμμάτα θα εγκριθούν τους επόμενους μερικούς μήνες και θέλουμε τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να ξεκινήσουν την υλοποίηση άμεσα ε, στη συνέχεια. Και όπως ε, ξέρετε υπάρχει Κάποια προβλήματα ε, είναι πιο επίγοντα. Αυτά που έχουν να κάνουν με την προβολία απασχόλησης των νέων. Υπάρχει μια ιδιαίτερη πίεση σε αυτά να ξεκινήσουν να λειτουργούν. Και εάν δεν ξεκινήσει θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. Thank you. There are no other comments. So the I, uh, oh, sorry. Still would like to ask the rapporteurs if there is. Να ζητήσουμε από τους ε, εισηγητές. Και μια τελευταία παρατήρηση. Οι σκιώδεις εισηγητές έχουν συζητήσει σε τόσους πολλούς τριμερείς διαλόγους και συζητήσει και εγκρίνει το κανονισμό τόσε πολλέ φορές. Θα θέλαμε να το, είχαμε, να το είχαμε ολοκληρώσει προηγουμένως, αλλά λόγω του Συμβουλίου δεν μπορέσαμε. Τέλος πάντων, πριν από το τέλος του προηγούμενου έτους, καταφέραμε να συμφωνήσουμε ε, στο βασικό, στο κανονισμό, το οποίο ήταν, είχε και μεγάλη σημασία για τα λειτουργικά προγράμματα. Απλώ σα θυμίζω ότι τα θέματα τα οποία αφορούν άμεσα τα λειτουργικά προγράμματα και τι εταιρικέ συμφωνίε. Υπό Κυπριακή Προεδρία είχαμε, ε, είχαμε κάνει τη διαβούλευση και είχαμε βρει μια βάση για την επεξεργασία των λειτουργικών προγραμμάτων η οποία υφίσταται. Δεν είναι λοιπόν σωστό ε, ότι οι περιφέρειες δεν είναι, δεν είναι πρόθυμες να προχωρήσουν με τα λειτουργικά τους προγράμματα. Ίσα ίσα ορισμένες περιφέρειες αρκετές ήδη ολοκληρώνουν τον προγραμματισμό των λειτουργικών προγραμμάτων και εγώ ως κοινοβούλιο δεν θέλω ουδόλως να δώσω το μήνυμα λίγο πριν από τις ευρωεκλογές ότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε επί αυτών των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων. Εγώ πιστεύω ότι αυτά που είπε η Κομισιόν μπορούμε να τα είναι απολύτως ε, σωστά και επιβεβαιώσιμα και δεν νομίζω ότι θα... Ε, είναι σε κάποιο από τον τομέα της αλληλείας ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώσει ή να απαντήσει 120 ερωτήσεις πιστεύω ότι αν καθυστερήσουμε για τον επόμενο έτος θα δώσουμε έναν τελώς λάθος μήνυμα και πιστεύω ότι το, όλη η ενημέρωση, όλες οι πληροφορίες υπήρχαν εξ αρχής Τώρα, εάν η αλία μας έκαιγε τόσο πολύ εξ αρχής, δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν είναι και δική μας ευθύνη. Εμάς ε, ο ρόλος μας ήταν να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη πρόταση και να ξεκινήσουμε φέτος με την εργασία αυτών των προγραμμάτων, με την υλοποίηση. Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Δύο θέματα θα ήθελα να θέσω. Τα έγγραφα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας έχουν γίνει δεκτά από το Συμβούλιο και δεν θα αλλάξουν. Θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση γι' αυτό. Εάν πράγματι ε, τα κείμενα αυτά είναι τα τελικά για το Συμβούλιο, Υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία δημιουργούν μια κάποια αβεβαιότητα και διαρωτώ με αν θα υπάρξει δυνατότητα περαιτέρω συζήτησης και αν πρέπει να προβλεφθεί μια χρονική προθεσμία. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν η συμφωνία την οποία είχαμε κάνει για τις κατεξουσιοδότηση πράξης προβλέπει ότι θα πρέπει στα πλαίσια της, ε, του ελέγχου της αξιολόγησης των επιδόσεων εμείς προβλέπουμε ίσως και κάποια διαφορετικά συστήματα. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι είτε εξάντε και στην περίπτωση που χρειαστεί να γίνουν κάποιες διορθώσεις ο τρόπος με τον οποίο ε, θα αλλάξει το σύστημα πρέπει να προβλεφθεί. Δεν μπορεί κανείς να αλλάζει αυθόρμητα οτιδήποτε. Είναι απαραίτητο λοιπόν αυτό για να μπορέσουμε μια, να έχουμε μια πιο ε, πράσινη ε, και μια πιο ευφυή απασχόληση για τους εργαζομένους. Όλα αυτά βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα συμπεριλάβει κανείς ε, σε ένα πρόγραμμα. Από την άλλη δεν πρέπει από την άλλη να έχουμε διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης κατά περίπτωση. Όταν λοιπόν τα προετοιμάζουμε αυτά θα πρέπει να κατανέμονται σωστά οι έλεγχοι και οι αρμοδιότητες ε, και κυρίως οι ευθύνες έτσι ώστε να μπορούν οι μικρομεσαίες να στηρίζονται και όχι να επιβαρύνονται μόνο γραφειοκρατικά. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα σχετικά με τις δικές μας διαχειριστικές αρχές. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι διαχειριστικές αυτές αρχές και πώς πρέπει ε, να εργάζονται στα διάφορα κράτη-μέλη. Πρέπει να μπορούν ανεμπόδιστα να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ότι τα πράγματα συστηματικά φαίνεται να μην διορθώνονται. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι μηχανισμούς θα χρησιμοποιούμε, να ξεκαθαρίσουμε το είδος των μηχανισμών που θα πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι ώστε να γίνονται οι διορθώσεις αυτές και οι έλεγχοι. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος των συγκεκριμένων κατεξουσιοδότηση πράξεων έρχονται ευρωεκλογές, η διαδικασία θα αργήσει να ολοκληρωθεί και αν κοιτάξει κανείς ε, το επίπεδο της λεπτομέρειας που έχουμε μπροστά μας, είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα αποφασιστούν αργότερα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε άλλωστε μία ακρόαση σχετική με το θέμα και θα τα ξαναθέσω όλα αυτά για να γίνω κατανοητός και για να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν ε, κάποιες συμβάσεις εταιρικών σχέσεων που έχουν ήδη κατατεθεί και δεν θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες καθυστερήσεις. Πρέπει να αποφύγουμε και στις περιπτώσεις αυτές και στις μελλοντικέ περιπτώσεις ε, να βάλουμε νέα εμπόδια, να ορθώσουμε νέα εμπόδια. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι για το διαφορετικό σύστημα το οποίο έχουμε μπροστά μας. Να μην κάνουμε τη ζωή των εμπλεκομένων δυσκολότερη. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο στον τομέα της εφαρμογής και να μην δημιουργήσουμε περισσότερα εμπόδια επαναλαμβάνει ο κύριος Ρόι. Και αν θέλει να σχολιάσει η Επιτροπή αυτά τα οποία είπαμε εδώ πρέπει να τα κάνει γρήγορα γιατί έχουμε λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες μάλλον μπροστά μας. Πρωτού κλείσω, Νίκολα, μήπως μπορείς να μας δώσεις συγκεκριμένες πληροφορίες για το Συμβούλιο. Ναι, Πρόεδρε. Είχαμε την ευκαιρία την περασμένη Παρασκευή να παρουσιάσουμε τις τρεις ε, κατεξουσιώδεις πράξεις στην ομάδα εργασίας και αυτό έδωσε την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να αντιδράσουν. Δεν ε, πρόκυψαν ε, μείζωνα θέματα. Γενικά υπήρξε στήριξη για τις κατεξουσιώδεις πράξεις και η Κομισιόν έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις ε, των συναντήσεων των εμπειρογνωμένων και άλλων κατών μελών που υπέδειξαν ότι ήταν έτοιμα να στηρίξουν. Δεν υπήρχε οποιαδήποτε αντίρρηση. Ευχαριστώ. Βίκτορ. Ναι, σε συντομία. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ανάγκη να παρατείνουμε τη συζήτηση ή τη διαμάχη εδώ, διότι Έχουμε συζητήσει εδώ και τόσους μήνες. Έχουμε συμφωνήσει πολύ περίπλοκα θέματα. Τώρα έχουμε πλησιάσει στην τελευταία περίπου συνάντηση της Ρέτζο. Αν δεν εγκρίνουμε τώρα τις κατεξουσδότητες πράξεις, τότε θα είναι πολύ αργά. Το επόμενο κοινοβούλιο θα αποτελείται από νεόφερτους, τουλάχιστον κατά το 50% και δεν είναι εύκολο να φανταστούμε πώς θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και σε συντομία με θέματα που, με τα οποία θα είναι λιγότερο εξοικειωμένοι. Είναι σημαντικό να εκπληρώσουμε το καθήκον μας τώρα, να εγκρίνουμε ε, ε, αυτό το θέμα και να δώσουμε αυτό το κληροδότημα στην επόμενη θητεία και να αφήσουμε τις περιφέρειες να αρχίσουν την υλοποίηση. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έχουμε τώρα την καταληκτική προθεσμία. Ιωαχήμ, είναι κάτι που θες να προσθέσεις. Τότε, να κάνουμε μια παρατήρηση. Εχθές πήραμε έναν κατάλογο κατά πόσο έχουν χρησιμοποιηθεί τα διαφορετικά τιμία από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που τα χρησιμοποίησαν κατά 50%, δηλαδή τα μέσα, τα κονδύλια που δικαιούνται εάν τώρα εφαρμόσουμε τους κανονισμούς ε, συν 2, συν 3, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπολογίσουμε κιόλα τα ποσοστά απορροφητικότητας. Ε, αυτή τη στιγμή τώρα βρίσκονται στη φάση της ε, περιγραφής της ουσίας των προτινομένων προγραμμάτων. Εδώ εμείς με τις πράξεις αυτές και τα παραδείγματα μιλάμε για τις τεχνικές πτυχές τι πρέπει να κάνουν και εδώ βλέπουμε ένα τεράστιο βάρος Πρέπει λοιπόν ε, να χρησιμοποιήσουμε την, αυτά που ξέρουμε από την εμπειρία μας. Και δεν είμαι βέβαιος ότι λόγω ορισμένων χαμηλών ε, ποσοστών απορροφητικότητας είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες υποδομές για τη βέλτιστη χρήση των κονδυλίων. Γι' αυτό ακριβώς και ανησυχώ για αυτά τα οποία ζητούνται εδώ να γίνουν. Η καταληκτική προθεσμία είναι 23 Μαρτίου. Το να ζητήσουμε παράταση δεν έχει νόημα, διότι δεν θα λύσει τα πράγματα. Αν θέλετε ε, να αντιταθείτε σε αυτή την πράξη, τότε μπορείτε να συντάξετε μια πρόταση ψηφίσματος. Ε, σας έχω πληροφορήσει για αυτά και εδώ θα ήθελα να κλείσω το θέμα αυτό και να επαναλάβω ότι η καταληκτική ημερομηνία 21η Μαρτίου και η Κωνσταντς ε, μίλησε πριν από τους άλλους ε, ομιλητές 12 ε, το μεσημέρι 21η Μαρτίου. Περνάμε τώρα στην επόμενη καταξιότητα της πράξη που σχετίζεται με ε, τους δικούς κανόνες σχετικά με τη μελετησομέτρια των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας. Επίσης, σε δύο μήνες έχουμε την προθεσμία, 4 Μαΐου δηλαδή. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να λάβει το λόγο. Η Σκιώδης, ε, η, ραπορτέρ, εισηγήτρια δεν είναι εδώ, η Σκιώδης. Έχουμε τη Μαρή Τερές, τον Φραντζέσκο Τάγγελης, τον Φρανσό Αλφονσί, τον κύριο Βλάσα, ανάμεσα στους σκιώδες ή να πάμε κατευθείαν στην Κομισιόν για τα σχόλια. Δεν υπάρχουν αγορητές. Νίκολας. Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος για τη συγκεκριμένη κατεξουσιοδότηση πράξη. Αυτό το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι συμβατό με τον κανονισμό ETC που ορίζει την επιλεξιμότητα και τους κανόνες της επιλεξιμότητας για τις κατηγορίες οι οποίες ε, συμμετέχουν εδώ. Καταρχάς υπάρχει υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρχεται εδώ και να ενημερώνει αναλυτικά. Κάτι το οποίο ήδη έχουμε κάνει εμείς από τις αρχές Μαρτίου. Το σκεπτικό μας είναι ότι ένας κοινός ε, κανόνας, ένα κοινό σύνολο κανόνων θα επιτρέψει την εφαρμογή του ETC ε και των προγραμμάτων του. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ το αντιφατικό, όλα βασίζονται στις ισχύουσες πρακτικές και τους ισχύοντες κανόνες και έχουν συζητηθεί επανειλημμένα στις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Ευχαριστώ. Η διαδικασία είναι η ίδια. Η προθεσμία είναι η 21η Μαρτίου, 12η Μεσημβρινή. Περνάμε στο 7 τώρα το οποίο είναι και αυτό μια κατεξουσιοδότηση πράξη, αφορά το ERDF. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής, ο Γιάνν Όλμπριχτ, θέλει κάτι να πει. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη πράξη, κατεξουσιοδότηση πράξη αφορά τις ε, κοινέ δραστηριότητες τις οποίες έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0,2 του ARDF το οποίο διανέμεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορά τις καινοτόμες πράξεις στον τομέα της αηφορίας ε, στην ανάπτυξη των πόλεων, των αστικών περιοχών. Εμείς ε, εργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις λεπτομέρειες. Η τελική διατύπωση είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να έχουμε να φτάσει στα κράτη-μέλη σύντομα. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Δεν θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση εκ νέου βέβαια, γιατί νομίζω ότι αυτή η κατεξουσιοδότηση πράξη έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει συγγνώμη να τεθεί σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατόν. Αν συμφωνήσουμε μόνο σε 5-6 μήνες, τότε θα ξεκινήσει τη δουλειά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση. Δεν θα χρειαστούν μόνο 6 μήνες, αλλά 8, 9, 10. Λοιπόν, δεν πρέπει να αργήσουμε άλλο. Αν πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο, ας μην το δεχτούμε. Όχι, δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, δεν είναι επικίνδυνο, είναι αποδεκτό αφορά τις καινοτόμες, καινοτομικές δράσεις. Έχουν γίνει συζητήσεις για κάποιες αλλαγές στους ορισμούς που χρησιμοποιούνται. Και εδώ στην ουσία αντιγράφουμε αυτά τα οποία λέει και ο δημοσιονομικός κανονισμός. Συνδέονται οι δύο κανονισμοί. Ορίζονται σωστά τα θέματα στα οποία θα υπάρξει δυνατότητα παρέμβασης. Δεν υπάρχει δυσκολία εδώ. Κάποιες παρατηρήσεις όμως θα ήθελα να κάνω, ίσως και κάποιες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη αφορά το ποσοστό συγχρηματοδότησης υπήρχε στην αρχική διατύπωση δεν υπάρχει τώρα. Ήταν Ποιο είναι αυτό το ποσοστό εν πάση περιπτώσει το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Στην αρχή υπήρχε η δυνατότητα απόκλησης και για τις μικρές χώρες. Η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει τώρα και υπάρχει θέμα ερμηνείας αν θέλετε ενός τμήματος του κανονισμού. Υπάρχει επίσης το θέμα της κατανομής σε ετήσια βάση. Μιλάμε για 330 εκατομμύρια που υπάρχουν για 7 χρόνια διαθέσιμα. Το θέμα είναι πώς θα διανεμηθεί στα μεμονωμένα ε, στα ετήσια χρονικά διαστήματα και επίσης ποιο θα είναι και το λειτουργικό κόστος. Υπάρχει επίσης και το θέμα του πάνελ των εμπειρογνωμόνων της ομάδας των εμπειρογνωμόνων. Ποια θα είναι τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία αυτής της ομάδας. Και τι θα γίνει επίσης και με τις προκηρύξεις. Πόσες τέτοιες προκηρύξεις θα υπάρξουν τα επόμενα 7 χρόνια λοιπόν. Αυτές είναι οι βασικές ερωτήσεις. Νομίζω ότι αφού ακούσω τις εξηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κάνω την τελική πρόταση ε, να προωθήσουμε το θέμα ως έχει. Σε ευχαριστώ πολύ Νίκολα. Ευχαριστώ ε, πρόεδρε. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό από την κανονισμό διότι εδώ αναφέρεται το πώς η Κομισιόν θα εφαρμόσει τις αστικές ε, και ανατομικές δράσεις. Ένας από τα, ένα από τα προϊόντα, από τα, από τα υποτελέσματα της ε, κατεξοδότησης πράξης ε, διαφέρει στον τρόπο εφαρμογής, δηλαδή πώς θα εκτελέσουμε αυτά τα προγράμματα και αναφέρεται κυρίως στο πεδίο ισχύως. Όπως είπε ο εισηγητής, ε, Χρησιμοποιούμε τώρα τη δυνατότητα κοινών διατάξεων, του κανονισμού κοινών διατάξεων, να εφαρμόσουμε ε, ε, έμεσες εκτελεστικές πράξεις και δίνουμε τη δυνατότητα διαχείρισης, η Κομισό δηλαδή μπορεί να δώσει ε, την διαχείριση σε φορείς εμπιστοσύνης. Ε, αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν περιλαμβάνονται πλέον στις, ε, στην εξουσιοδότηση πράξη η, τα ποσοστά στη χρηματοδότηση ή στοιχεία χρηματοδότησης καθόλου δεν υπάρχουν, διότι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν καλύπτεται από την εξουσιοδότηση, από το πηδέν ισχύω της εξουσιοδότησης. Και θα ασχοληθούμε, θα καλύψουμε τις χρηματοδοτικές πτυχές σύμφωνα με τον χρηματοδοτικό κανονισμό. Άρα λοιπόν τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν εδώ και μπορούν να τροποποιηθούν αυτές οι διατάξεις ε, ανάλογα με την φύση του κάθε αιτήματος και θα μπορούν ε, να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές ε, διατάξεις συγχρηματοδότησης κατά την πορεία της υλοποίησης. Ο λόγος για τον οποίο ζητούμε αυτή την παρέκκληση για τα μικρά κράτη-μέλη είναι ότι έχουμε χρησιμοποιήσει στο σχέδιο σύνταξης ε, ως ελάχιστο όριο κατοίκων τις 50.000 για τις περιφέρειες και τώρα χρησιμοποιούμε την προσέγγιση της Eurostat η οποία ορίζει ένα, μια αστική πόλη, μια πόλη ε, σύμφωνα με τον ορισμό και την ερμηνεία του ΟΣΑ και της Eurostat. Ε, τώρα, βλέποντας ε, την πρακτική εφαρμογή αυτού του ορισμού δεν δημιουργεί ανομαλίες ή στρεβλώσεις στα κράτη-μέλη. Αλλά ε, και η Μάλτα, ας πούμε, και η Λευκοσία καλύπτεται από τον ορισμό αυτό. Έχουμε λοιπόν βάσει της διατύπωσης των ορισμών αυτών τη δυνατότητα ομαδοποίησης ε, πόλεων όπου ο πληθυσμός είναι κάτω από 50.000 μπορούμε να ομαδοποιησουμε δυο 2-3 πόλεις μαζί μικρότερες ε, και να ε, τις ενοποιήσουμε για να μπορέσουμε να τις καλύψουμε με τα κριτήρια που σε σπίστηκαν. Δεν χρειάζεται τότε λοιπόν παρέκκληση και γι' αυτό δημιουργήθηκε μία συνέπεια στην προσέγγιση δεν έχουμε επιτέλθει σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα κριτήρια των ε, εμπειρογνωμόνων, ε, των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Δεν υπάρχει λόγος να ανακαλύπτονται από τις κατεξοδότητες ε, πράξεις, αλλά οι λεπτομέρειες θα τεθούν μεταξύ της συμφωνίας με την αρχή ανάθεσης και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια πολύ καλή βάση επιλογής. Μια πολύ καλή διαδικασία επιλογής και θα ενημερώνουμε βεβαίως το Κοινοβούλιο όσον αφορά την υλοποίηση αυτής της πράξης και θα ζητούμε την ε, συμβολή σας ε, όσον αφορά την κάλυψη των θεμάτων που εμπίπτουν σε αυτή την πράξη. Η Κορνέλια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν τι συμβαίνει με το, με το εξή σημείο. Λοιπόν, η Κομισιόν κάνει μια συμφωνία με τον φορέα ε, ανάθεσης και υπάρχουν και αυτές οι ομάδες εμπειρογνωμόνων και αυτό πρέπει να συζητηθεί με την Κομισιόν. είπετε τώρα ότι αυτοί οι εμπειρογνώμονες, αυτοί οι φορείς εμπειρογνωμόνων δεν θέλετε να ε, αναμειχθείτε, δεν χρειάζεται να καθορίσετε όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχουν προτάσεις και ένας κατάλογος εμπειρογνωμόνων που θα ε, τον μελετήσει η Κομισιόν. Ε, στον κατάλογο αυτό θα υπάρχουν και οι φορείς, οι εγκεκριμένοι φορείς, ε, θα υπάρχει ένας τελικός κατάλογος μεταξύ των φορέων των εγκεκριμένων ή φορέων εμπιστοσύνης και των ε, εμπειρογνωμόνων. Με ενδιαφέρει λοιπόν ποια είναι η διαδικασία πριν από την έγκριση ε, μιας αίτησης μεταξύ της αξιολόγησης από την Κομισιόν και της συμβολής των εμπειρογνωμόνων πριν γίνει η ανάθεση στους φορείς. Α, συνεχίζει η ομιλήτρια και στη συγχρηματοδότηση λέτε ότι θα πρέπει να προσαρμόζεται, να υπάρχει ένα μοντέλο ανάλογα με την, ε, της, ε, με την διαδικασία διαγωνισμού προς ανάθεση. Δηλαδή υπάρχει κάποια ευελιξία εδώ από ό,τι βλέπω στη χρηματοδότηση. Εάν η χρηματοδότηση είναι πολύ χαμηλή, ε, μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πράξη και να καλύπτει μια κοινότητα. Υπάρχουν τι όρια υπάρχουν αριθμητικά, πώς ερμηνεύεται εν πάση περιπτώσει αυτά τα στοιχεία της κοινότητος, διότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τους κατοίκους. Νίκολας. Ευχαριστώ για τις ε, επιπρόσθετες ερωτήσεις. Το κλειδί για την Κομισιόν ήταν να έχουμε την εποπτεία στη διαδικασία επιλογής. Αυτή ήταν η μεγάλη απόφαση, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι καινοτόμες ε, πράξεις αστικές ε, παραδίδουν ενδιαφέροντα προγράμματα και ότι κερδίζουμε κάτι από αυτή τη διαδικασία. Αυτό λοιπόν καθορίσαμε μια διαδικασία όπου ο φορέας θα κάνει τη δουλειά στην προκήρυξη και την επιλογή της διαδικασίας. Θα υπάρχει ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων με την Προεδρία της Κομισιόν και ότι η Κομισιόν θα αναθεωρήσει όλες τις προτάσεις και θα κάνει συστάσεις και η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον φορέα σε συμφωνία με την Κομισιόν. Δίνει λοιπόν άμεση εμπλοκή στην Κομισιόν στην τελική διαδικασία Βεβαίω, με βάση τις συστάσεις που προέρχονται από το πάνελ των εμπειρογνωμόνων. Θέλουμε να υπάρχει μια διαφανής διαδικασία όσο το δυνατόν, να έχουμε ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων με ε, πλατιά εμπειρία, έτσι ώστε να έχουμε γερές συστάσεις, αλλά η Κομισιόν θέλει να διασφαλίσει ότι αυτό το μέσο παραδίδει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Επίσης, δημιουργούμε εδώ ένα πλαίσιο, αλλά δεν είναι μια διαδικασία εφάπαξ. Θα έχουμε μια σειρά από τέτοιες διαδικασίες και θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε από τις εμπειρίες και να ρυθμίσουμε τελικά και να κάνουμε τις τελικές ρυθμίσεις. Και αν ε, είναι απαραίτητο να έχουμε και οποιαδήποτε τροπολογία στην ε, ε, στην πράξη. Δηλαδή αν κάτι πρέπει να ενισχυθεί, αν κάτι λείπει, ε, δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα, στη συγχρηματοδότηση. Όλα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το δημοσιονομικό κανονισμό. Ε, αλλά Ε, να μην έχουμε πολύ ψηλέ απαιτήσει. Δέχομαι αυτό το σημείο. Θα πρέπει να έχει επιτυχία. Δεν έχει νόημα να ξεκινήσουμε με μια απέτηση προ... Ε, ε, συγχρηματοδότησης που δεν θα είναι δυνατόν να την καλύψουν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Θα πρέπει να προβλέψουμε το επίπεδο συγχρηματοδότησης να είναι επαρκές για να έχει επιτυχία αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια Γιάννα, θα ήθελες να κάνεις ένα τελικό σχόλιο. Όχι κάτι. Άρα, ίδια διαδικασία ακολουθείται. 21η Μαρτίου είναι η προθεσμία, 12η μεσημβρινή, για όλους όσους θέλουν να παρουσιάσουν ένα σχέδιο πρότασης ε, με τις αντιρρήσεις τους. Εδώ κλείνει αυτό το σημείο. Θα συναντηθούμε στις 3 η ώρα. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Κεφαλαίων από τη Ρουμανία και θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Πέρα ε, της συνεδρίας.